Καλώ eh, Καλώς ήρθατε στην ε, σημερινή ακρόαση που έχει θέμα την κατάσταση των γυναικών στο πόλεμο. Η ακρόαση αυτή αποτελεί μέρος ε, της εργασίας ε, για μια έκθεση πρωτοβουλία στο θέμα για την οποία είναι υπεύθυνη η κυρία Νικολάη. βλέπω ότι μας περιμένει ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Ε, εν μέρη λόγω του θέματος ε, της ημέρας αυτής που είναι τόσο σημαντικό και εν μέρη λόγω της προοπτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ε, τη σχέση δηλαδή ανάμεσα ε, το, το θέμα της ε, ε, εξωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης λόγω των ομιλητών, των μας σήμερα που έχουν πολλή εμπειρία και πολλές γνώσεις στον τομέα αυτών. Θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το απόγευμα που θα περάσουμε μαζί. Η σημερινή ακρόαση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο θα είναι μια συζήτηση πάνελ με θέμα το ρόλο των γυναικών ε, στις ε, στρατιωτικές δομές ε, στα πλαίσια των πρωτοβουλειών για ειρήνη και ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του προγράμματος και το δεύτερο είναι συζήτηση σε πάνελ πάλι για το θέμα οι συνέπειες των συγκρούσεων στις γυναίκες. Και Πρωτού να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα ε, να σας πω το εξής για το θέμα της ημέρας. Το να ζήσει κανείς έναν πόλεμο είναι μια από τι χειρότερε καταστάσει που μπορεί να ζητήσει κανείς ε, και για άντρες και για γυναίκες. Το να ζήσει κανείς ε, την βία, τον τρόμο, Το να δει κανείς ε, πώς παιδιά, συγγενείς, φίλοι χάνονται, πώς διαλύεται όλο ο ιστός της κοινωνίας. Και βλέπουμε ότι ε, οι γυναίκες πλήττονται ακόμα περισσότερο από τη βία λόγω του φίλου τους. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταστάσεις που μπορεί να ζήσει κανείς. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν οι καταστάσεις αυτές. Ξέρουμε ότι οι πόλεμοι Ε, είναι καταστάσεις που πολύ δύσκολο είναι να λυθούν. Και οι, ε, οι συνθήκες ε, υπό τις οποίες αναγκάζονται να ζουν γυναίκες ε, στις καταστάσεις αυτές είναι μια επιπλέον πτυχή στην, στις καταστάσεις αυτές. Αλλά η συνείδηση η προσπάθεια να βρεθούν λύσεις, να υπάρξει επικοδομητικός διάλογος, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικές στα διάφορα επίπεδα. Μιλάμε εδώ για το διεθνές επίπεδο, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην εξέβρεση λύσεων για το μέλλον. Διότι όλοι συμφωνούν ότι δεν θέλουμε οι καταστάσεις αυτές να αποτελούν πραγματικότητα για τους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ε, το σημερινό απόγευμα και τη δουλειά της ε, κυρίας ε, Νικολάη που έχει σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας της, θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ένα μέρος της προσπάθειας εξέβρισης λύσεων. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην σημερινή ακρόση και δίνω το λόγο στην κυρία Νικολάη που είναι υπεύθυνη εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που λαμβάνω μέρος σε αυτή τη δημόσια κρόαση γιατί πιστεύω ότι το αντικείμενο αυτής της ακρόασης είναι ένα θέμα που μας δείχνει τα όρια του πολιτισμού μας στον 21ο αιώνα και γιατί μιλάω για όρια. Θα μιλήσω για τα όρια αυτά όχι μόνο ως μέλος της Επιτροπής Γυναικών, αλλά και ως Αντιπρόεδρος Υποεπιτροπής για την Άμυνα. Η βία εις βάρος των γυναικών ήταν Πραγματικά η αποδός της ανθρώπινης ναυσότητας που αποκαλείται πόλεμος, ακόμη και αν μιλάμε για τον κλασικό γνωστό πόλεμο από την αρχαιότητα, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι είχαμε ανέκαθεν πολέμους, πόλεμοι και βιαιότητες στις βάρος των γυναικών αναφέρονται ακόμη και στη βίβλο, αλλά στη περίπτωση της θρησκείας παρόλο που δεν δεχόμαστε την εξήγηση, υπάρχει μία εξήγηση. Αλλά όλοι ε, προσπαθούν να βρουν μία εξήγηση μέσω της θρησκείας για τέτοιου είδους βιοπραγίες. Και αυτές οι εξηγήσεις και αυτές οι δικαιολογίες συνεχίστηκαν παρά την ε, περαιτέρω ανάπτυξη και εκλέπτηση, εξήτηση του πολιτισμού. Θυμόμαστε τα πρόσφατα γεγονότα της Λιβύης. Τα συμβάντα στη Λιβύη, αυτό που συμβαίνει σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε μια πολιτισμένη κοινωνία με κανόνες, καταδεικνύουν ότι τέτοιου είδους βαναυσότητες, φρικαλαιότητες ε, δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό. Μπορεί να χρησιμοποιούνται ως μοχλός από τον πολιτισμό, αλλά δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από τα όρια του πολιτισμού. Γινόμαστε σήμερα μάρτυρες σε πολλά μέρη του κόσμου, ενός διαφορετικού είδους κοινωνίες, γινόμαστε μάρτυρες πολλών φαινομένων επιθετικότητας εις βάρος των γυναικών. Και ακόμη και αν ο βιασμός έχει αναγνωριστεί ως έγκλημα πολέμου, δυστυχώς τα διεθνή συστήματα ενώμης τάξης δεν κατάφεραν να προλάβουν ή να τιμωρήσουν τους αυτούργους. Γιατί αυτά τα δύο σημεία θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου. Μία πρόληψη αποτελεσματική, οργανωμένη, αλλά και μία καταστολή, μία τιμωρία, μία επιβολή ποινών που θα είναι ε, σωστή και αποτελεσματική. Δυστυχώς και αυτά τα δύο στοιχεία λείπουν, και η πρόληψη και η τιμωρία. Και δυστυχώς ε, δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη. Στην Ευρώπη, γιατί εγώ οφείλω να περιοριστώ στην κατάσταση αυτή της Ευρώπης, θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες γιατί βρισκόμαστε ήδη στα άκρα μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Και θα ήταν σκόπιμο να έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό, ήδη από τώρα και να συμπεριλάβουμε και αυτό το ζήτημα στην κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας, στην ΕΠΑ. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο και μπορούμε να θεσπίσουμε κοινούς κανόνες, κοινέ προδιαγραφές και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και να λάβουν υπόψη στις πολιτικές τους τη βιοπραγία εις βάρος των γυναικών. Έχουμε πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ και πολλές σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες και μάλιστα σήμερα έχουμε και μία επίτροπο αρμόδια για το θέμα αυτό στον ΟΗΕ ή μάλλον μια υπάτη αρμοστή. Υπάρχει, θεσμοποιηθεί λοιπόν αυτή η ειδική αρμοδιότητα στην υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ. Αλλά η κατάσταση αυτή θα παραμείνει αναποτελεσματική και θα έχει απλώς αξία διακηρυκτική αν δεν συνεργαστούμε εμπράκτος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εμπλακεί ενεργά και η Ευρώπη στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσουμε το θέμα. Και δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να προσεγγίσουμε ταυτόχρονα πολλά μέτωπα. Χαίρομαι που έχουμε προσκαλέσει και εμπειρογνώμονες στη δημόσια κρόαση και καλύτερα θα είναι να τους δώσουμε το λόγο και να υποφεληθούμε από την παρουσία τους και την, τις γνώσεις τους. Γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ εδώ, για να αξιοποιήσω και να διδαχτώ από τις γνώσεις, γιατί ωραία είναι να διαβάζουμε και να ακούμε ορισμένα πράγματα, αλλά το καλύτερο είναι οι έμπρακτες γνώσεις, η πραγματογνωμοσύνη, η εμπειρογνωμοσύνη. Αυτές είναι που θα δώσουν και μια νέα πτυχή και μια νέα αξία στην προσέγγιση του θέματος αυτό. Και μάλιστα θα μας υποδείξουν και κάποιες λύσεις. Αυτά περιμένουμε από την έκθεση αυτή. Περιμένουμε πρόταση για κάποιους κοινού μηχανισμούς, μηχανισμούς συνεργασίας, που θα είναι και αποτελεσματικοί, προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών στις, ε, σε εμπόλεμες καταστάσεις. Γιατί σήμερα έχουμε πολλούς και διαφορετικούς πολέμους. Έχουμε... Η κλασική μορφή του πολέμου, όπως τη γνωρίζουμε από την ιστορία, έχει... είναι πια ξεπερασμένη. Πολλοί και διαφορετικοί πόλεμοι λαμβάνουν χώρα σήμερα, που είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από την κλασική μορφή του πολέμου, γιατί δυστυχώς οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν υπακούουν σε κανένα κανόνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευελπιστώ, είμαι σχεδόν βέβαιη ότι θα έχουμε πολύ καρποφόρα συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νικολάη. Θα χαρώ πολύ τώρα να καλωσορίσω την Ελίσα Πέτρεένα από τη Φιλανδία που είναι πρόεδρος του Συμβουλίου ε, για τα θύματα του ε, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ε, σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσα να μιλήσω και σου ειδικά. Υπάρχει διερμηνία από ό,τι βλέπω, αλλά έχω ετοιμάσει την ομιλία μου στα αγγλικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ συμμετείχα στην ηγεσία, υπήρξε υπουργό, υπήρξε και ευρωβουλευτής εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, συμμετείχα και στην ε, ε, αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι έμαθα πολύ περισσότερα για το όλο θέμα τα τελευταία 10-15 χρόνια ε, που ασχολούμαι πλέον με τα θύματα των ε, σειράξεων, διότι εκεί είναι που μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ιδίω τώρα που έχει αλλάξει εντελώ η φύση των σειράξεων. Δεν πρόκειται πλέον για σύριαξη μεταξύ δύο ανεξαρτήτων χωρών, δεν είναι ε, πόλεμος για τα σύνορα ή για οποιαδήποτε άλλη διαμάχη μεταξύ τους. Πρόκειται για έναν εσωτερικό πόλεμο, ένα παιχνίδι εξουσία, ένα οικονομικό, πολιτικό πρόβλημα, μπορεί να είναι τα διαμάντια, τα διάφορα μέταλλα, και όλοι οι φυσικοί πόροι και το θέμα της ανθρώπινης εξουσίας αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για αυτές τις ε, σημερινές ε, σειράξεις. Και δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα θύματα είναι πάντα οι πολίτες, ιδίως οι γυναίκες σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Οι πιο ευάλωτες ομάδες δηλαδή. Και επιπλέον Μία από τις τακτικές του πολέμου, ε, για να αποτελεί και το κερασάκι στην, ε, είναι ο βιασμός. Είναι μια πολύ επιτυχημένη τακτική, διότι όταν βιάζεται κάποιος, βιάζεται η όλη του οικογένεια, το ίδιο χωριό, ε, όλος ο περίγυρός του. Πρόκειται για κάτι λοιπόν το οποίο είναι πονίδιστο. Και ε, να σας υπενθυμίσω ότι δεν βιάζονται μόνο γυναίκες και νεαρά κορίτσια, αλλά και άνδρες. Και κατά κάποιο τρόπο τα θύματα τα οποία συνάντησα ε, που είναι άντρες είναι σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση διότι ε, όταν βιάζεται ένας άνδρας ε, χάνει και την περηφάνειά του, την αξιοπρέπειά του όλα αυτά χάνονται με το βιασμό θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι οποιοδήποτε αποτελεί στόχο σεξουαλικής βίας θα πρέπει να καταδικάζουμε το φαινόμενο Ο πόλεμος και ο βιασμός είναι αλληλένδετοι. Διότι πολλές φορές ε, μου είπαν ότι θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ε, τις τοπικές γλώσσες, διότι πολλές γλώσσες δεν έχουν τον όρο βιασμός, αλλά μετά από ένα πόλεμο σε μια περιοχή υπάρχει πλέον όρος. Χρειάστηκε να δημιουργηθεί δηλαδή ο όρος στην τοπική γλώσσα πολλές φορές, έτσι μου λένε. Το ψήφισμα 2025 των Εθνών ε, πρόκειται να αφορά την πρόληψη και τη συμμετοχή των γυναικών, ιδίω τη συμμετοχή των γυναικών ως συμμετέχοντες στην ειρήνη και την ασφάλεια. Και να μην θεωρούμε τις γυναίκες αποκλειστικώς και μόνον θύματα. Όπως ε, μου είπαν ε, πολλές φορές στις χώρες στις οποίες επισκέπτομαι, επειδή συμμετέχω και ως ε, ε, μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μου είπαν ότι δεν θέλουμε να αποκαλούμαστε θύματα, αλλά θέλουμε να αποκαλούμαστε επιζώντες. Αυτές οι γυναίκες είναι ισχυρές, διότι επέζησαν, θέλουν να ε, δημιουργήσουν και προσβλέπουν σε ένα καλύτερο μέλος για τις χώρες τους. Και αυτό δε, σημαίνει ότι δεν θέλουν να θεωρούνται θύματα, διότι ένα θύμα είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε μειονεκτικό. Μετά από το 2025 και όλα τα σχετικά ψηφίσματα που είχαμε σε 10 χρόνια, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε κάτι ε, άλλο πέραν από νέα ψηφίσματα. Το 1820, το 1880, το 1889 και ούτω καθεξής. Και σε κάποιο βαθμό όλα αυτά τα ψηφίσματα επιδεινώνουν την κατάσταση των γυναικών, αν μου επιτρέπετε να σας το πω αυτό. Διότι οι γυναίκες θεωρούνται θύματα και δεν θεωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και οι, οποίοι θα, οι οποίες θα πρέπει να εμπλέκονται στην όλη διαδικασία και σε ηγετικέ θέσεις και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ανταυτού τις κάνουμε θύματα. Και βεβαίω αυτό δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ε, τις βοηθήσουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τουλάχιστον κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να πω ότι η διεθνή κοινότητα δεν υπήρξε ιδιαίτερα στεναρή, δεν αποτέλεσε πρότυπο, διότι δεν αναλαμβάνουν γυναίκες την γεννησία ειρηνευτικών αποστολών και δεν αναλαμβάνουν γυναίκες ως εκπρόσωποι. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η, για τις γυναίκες, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κάτι φρικτό. Πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να υπάρξει μια γυναίκα εκπρόσωπος και ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε ε, να διοριστεί η επόμενη γυναίκα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σύντομα. Και μην μου πείτε ότι ψάχνουμε αξίες και προσόντα και δεν ασχολούμαστε με το φύλλο. Διότι αυτό ε, θα σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα για να αναλάβουν ως επικεφαλής ε, μιας αποστολής ή να είναι, είπατε, εκπρόσωποι κάπου. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο εδώ ε, και πιέζουμε επί του θέματος. Διότι όταν κάποιος έχει έναν ηγετικό ρόλο στη διεθνή κοινότητα, κατά κάποιο τρόπο θεωρείται πρότυπο. Εάν μπορεί μια γυναίκα λοιπόν να ε, έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο, οι υπόλοιποι θεωρούν ότι και εμείς μπορούμε. Και όλο αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι και οι συγκρούσεις αυτή τη στιγμή είναι όπως είναι. Η διεθνής αστυνομία, η πολιτική αστυνομία, οι ειρηνευτικές δυνάμεις ε, πάντα περιλαμβάνουν ε, στις περιφέρειες και τις γυναίκες, διότι επειδή τα εγκλήματα είναι έτσι όπως είναι και επειδή πολύ συχνά η οικογενειακή βία έρχεται ως συνέπεια της βίας του πολέμου και του πολέμου. Για πολλές γυναίκες είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να αποτανθούν σε έναν άντρα και να καταγγείλουν ότι αποτέλεσαν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή ε, θύμα οικογενειακής βίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να στραφούν σε μια γυναίκα, αστυνομικό ή ε, στρατιώτη για να της πούν τι ακριβώς συνέβη. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό και με ενοχλούν οι μεγάλες ειρηνευτικές αποστολές ε, όπου ε, έχουμε στις ειρηνευτικές δυνάμεις ανθρώπους από το Πακιστάν που δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά δεν περιλαμβάνονται καθόλου γυναίκες στα στρατεύματά τους. Και αυτό είναι ε, πολύ δυσάρεστο όταν υπάρχουν εκατοντάδες στρατιώτες και δεν υπάρχει καμία γυναίκα που θα μπορούσε να συνδράμει τις γυναίκες επιτόπου. Οι γυναίκε όμω, οι οποίε συμμετέχουν στι ειρηνευτικέ αποστολέ και στι αστυνομικέ δυνάμει, θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση προηγουμένω. και αυτό θα πρέπει να το απαιτούμε. Ε, δεν σημαίνει ότι θα πάει μια γυναίκα, θα λάβει μία ώρα εκπαίδευση και θα του πείτε ότι κοιτάξτε να δείτε θα βιάζονται και οι γυναίκε και δεν θα πρέπει να τι βιάζετε. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επιμόρφωση, να γνωρίζουν τον πολιτισμό, την οτροπία, τι παραδόσεις και τη συμπεριφορά αυτών των χωρών στις οποίες ε, θα μεταβούν. Και αυτό φυσικά έχει σημασία. Ένα από τα προβλήματα που διαπίστωσα στις αποστολές μου στην Αφρική ιδίω, αλλά και σε άλλες περιοχές είναι ότι ο πολιτισμός και η νοοτροπία είναι τόσο πολύ υπέρ των ανδρών και των συζύγων όπου σε χώρες όπως την Ουγκάντα ή και σε άλλες αφρικανικές χώρες, όταν μια γυναίκα είναι σύζυγος και βιάζεται στη διάρκεια της νύχτας από 10 στρατιώτες, για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να τους αναγνωρίσει, φορούν ε, ε, μάσκες, κάποια μεταμφίεση, τότε ο σύζυγος απορρίπτει τη γυναίκα και όλα τα παιδιά διότι θεωρεί ότι είναι άπιστη, γιατί κοιμήθηκε με άλλους άνδρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το αναγνωρίζει η τοπική κουλτούρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ε, η ανδρική περηφάνεια δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι υπήρξε άπιστη η γυναίκα του και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Το συζήτησα και με τη Μάργκοτ Μάλστρομ, επανειλημμένος, αλλά δεν ε, εισακουγόμαστε. Θα πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη προσπάθεια ώστε οι άνδρες να συνταχθούν μαζί μας και να συνεργαστούν μαζί μας, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας ζητήσω. Ε, το ζητώ και από τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας μου και πάντα το επενθυμίζω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική ατζέντα για θέματα φύλου και σεξουαλικής βίας σε, όλα, σε όλες τις πολιτικές ασφαλείας και άμυνας, σε όλες τις πτυχές. Όταν συζητάμε ειρηνευτικέ συμφωνίες θα πρέπει να μην λησμονούμε, να περιλαμβάνονται στι ε, συζητήσει και το θέμα τη ενημέρωση σε θέματα φύλου και της ε, συμπερίληψη των γυναικών ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρέπει να θεωρείται ένα εξωρετικό ζήτημα και να το εξετάσουμε μεμονωμένα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα διέπει όλα τα ζητήματα τα οποία συζητώνται. Γιατί απαιτούνται όμως οι γυναίκες ε, στις στρατιωτικές δομές, γιατί είναι απαραίτητες ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Καταρχάς γνωρίζουν πολλά για τα πρακτικά ζητήματα, αλλά επιπλέον γνωρίζουν και πώς ε, είναι οι δομές όταν υπάρχει διαπραγμάτευση για την ειρήνη. Υπάρχει για παράδειγμα ζήτηση για τιμωρησία, για αμνηστία και έχω δει πολλές περιπτώσεις τις οποίες στιγματοποιούνται τα θύματα, απομακρύνονται από την κοινότητα, από το χωριό τους, ενώ οι ε, βιαστές ε, απολαμβάνουν αμνηστίας και συνεχίζουν να ζουν ε, μια χαρά στην ίδια την κοινότητα. Ακόμα και τα ε, ε, παιδιά αντιμετωπίζονται με άσχημο τρόπο. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίξουν με άλλα παιδιά στο χωριό γιατί ε, ο πατέρας του θεωρείται ο εχθρός, αλλά ο πατέρας είναι αυτός που έχει την εξουσία. Η γυναίκα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να θίξει και αυτά τα θέματα και να ζητήσει, να πιέσει, να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία. Πριν από μερικέ εβδομάδε πήγα και πάλι στην αγαπημένη μου Βοσνία Ερζεγοβίνη, μίλησα με γυναίκες από τη Σρεμπρένιτσα στο εργαστήριο DNA, όπου είχαμε 3.500 ε, πακέτα τα οποία ακόμα περιμένουν αναγνώριση. Μίλησα με γυναίκες και όλες μου είπαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς να αποδοθεί δικαιοσύνη. ο Ομπάμα κατάφερε να πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάνταν, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει τον Μλάντιτς. Αυτή τη στιγμή ε, και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ε, έχω μόνο ένα λεπτό, θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Όπως σας είπα, δεν μπορούμε να περιθωριοποιηθούμε. Αναφερόμαστε στα δικαιώματα των γυναικών και στην κατάσταση των γυναικών. Ήταν σφάλμα κατά την άποψή μου οι γυναίκες στα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν το, την ονομασία γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών, διότι πάλι μας αντιμετωπίζουν στην απομόνηση. Δεν υπάρχει αντίστοιχο ε, θέμα όπως άνδρες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ σημαντικό οι άνδρες και οι γυναίκες να συνεργάζονται από κοινού και να προσπαθούν να επιτύχουν αποτελέσματα και να σέβονται τις γυναίκες όπως θα έπρεπε. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θύματα, αλλά ως επιζώντες, ως ε, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας τους μέσω δέσμευσης και συμμετοχής τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες αυτές ε, πληροφορίες. Ε, σημειώνουμε αυτά που είπατε και θα τα σκεφτούμε και θα ήθελα ιδιαίτερα να, σημειώσω, να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να ξεφύγουμε από τον ρόλο του θύματος ε, των γυναικών, ε, να δούμε τις γυναίκες ως ε, ε, επιζώντες που τα καταφέρνουν καλά, που, διότι έτσι είναι στην πραγματικότητα. Αυτός ε, είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ θερμά και θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την Μάιμπριτ Τεωρίν από τη Σουηδία. που ε, έχει ε, πολύ πείρα ως ε, πρέσβησε για, για τον αφοπλισμό, έχει πολύ πείρα από τις εργασίες στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συγκεκριμένη μας Επιτροπή. Σας καλωσορίζω θερμά λοιπόν και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι πάλι εδώ στην Επιτροπή Γυναικών και ιδιαίτερα χαίρομαι που ε, θίγεται το θέμα αυτό. Και εγώ θα μιλήσω αγγλικά. Το μισό του παραδείσου ε, το στηρίζουν οι γυναίκες. Αλλά στις ε, ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ασφαλείας δεν είναι παρούσα η γυναίκα. Και παραθέτω και στο παρελθόν ε, ε, και τώρα... Ε, συγχωρούσαμε και καταλαβαίναμε αυτά που κάνανε οι άντρες ε, και ε, καταλαβαίναμε και το κόλπο σας. Μέναμε εδώ και ακούγαμε ότι είχατε κάνει κάτι ανόητο και ρωτούσαμε πώς τα καταφέρατε με την Ειρηνευτική Συμφωνία. Συμφωνήσατε σχετικά με την ανακοίνωση που θα πρέπει να σκαλιστεί σε λίθο ο άντρας απαντάει «Μην ανακατεύεσαι, άφησε με ήσυχο». Ε, και εγώ σώπασα. Τα λόγια αυτά είναι από τη Λυσιστράτη. Ε, στο έργο του Αριστοφάνη 411 χρόνια πριν ε, π.Χ. Θα μπορούσαν όμως κάλλιστα τα ίδια να τα πούνε οι γυναίκες σήμερα. Από την εποχή της Λυσιστράτης οι γυναίκες στις γυναίκες ε, λένε να μην ε, ασχολούνται με τους πολέμους των ανδρών ε, και τις ειρηνευτικές διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη εάν δεν επιτρέπεται στο μισό της ανθρωπότητας να συμμετέσχει στην επίλυση των κρίσεων και στη διαπραγματεύση της ειρήνης. Ακόμα και σήμερα ακόμα και αν έχουμε περισσότερη ισότητα σε άλλους τομείς, η κατάσταση είναι ίδια που ίσχυε για τη Λυσιστράτη και τις αδερφές της. Εμ αλλά το μισό του παραδείσου το στηρίζουν οι γυναίκες και γι' αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν ε, στις εργασίες αυτές. Ε, στις ε, διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στο Τατζικιστάν μόνο μία γυναίκα ήταν μεταξύ των 26 εκπροσώπων παρότι ο πόλεμος είχε χειρέψει 25.000 γυναίκες. Στην Αρούσα, στις διαπραγματεύσεις για τον Μπουρούντι, μόνο δύο από τους 125 εκπροσώπους ήταν γυναίκες και ε, στην ε, Σιέρα Λεόνε, παρά τις ε, πολύ βάρβαρες επιθέσεις που είχαν γίνει κατά γυναικών και κοριτσιών, οι διαπραγματεύσεις αυτές έκλειναν τα μάτια μπροστά στις, στα δικαιώματα των γυναικών και τις προτεραιότητες τους. Και τι εικόνα έχουν σήμερα οι νευτικές διαδικασίες, οι ίδιοι, άντρε, οι ίδιοι που ξεκινούν τον πόλεμο, μετά διαπραγματεύονται για την ειρήνη. Καμία γυναίκα δεν είναι παρούσα. Ε, έχει έρθει η ώρα να δώσουμε τέλος ε, στην ε, μεγάλη σιωπή, όπως είπε χθες η Κλόντια Μεζία Ντούκ από την Κολομβία σε μια συνάντηση στη Στοκχόλμη. Εδώ και 50 χρόνια γίνεται πόλεμος στην Κολομβία με 5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, εκ των οποίων το 80% είναι γυναίκες. Είπε ότι κάθε ώρα δύο γυναίκες πέφτουν θύμα σεξουαλικής βίας και το 84% από αυτές είναι ε, ακόμα παιδιά ή ε, νέες κοπέλες. Ε, η σεξουαλική βία ασκείται και από τις στρατιωτικές και από τις παραστρατιωτικές ομάδες ε, και από 51.616 τέτοιε πράξει, μόνο ε, τι 42 ε, παραδέχτηκαν οι δράστε και πολύ λίγε ε, έφτασαν στα δικαστήρια, ενώ ακόμα, ακόμα λιγότερες ήταν οι καταδίκες τελικά. Αυτή είναι η Κολομβία σήμερα. Και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει. Καμία γυναίκα δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ειρήνης που έδωσαν τέλο τον πόλεμο στην Βοσνία, παρά το γεγονό ότι όλο ο κόσμο ήξερε για του βιασμού που είχαν γίνει κατά γυναικών. Ε, ακόμα και τώρα δεν είναι καλύτερα ε, τα πράγματα. Στην ε, οργάνωση Operation 1325 που είναι μια ένωση πέντε ενώσεων ειρήνης και γυναικών στη Σουηδία το το 2008 ε, εξετάσαμε πόσες ε, γυναίκες ε, συμμετείχαν στις ειρηνευτικές αποστολές, όχι τις στρατιωτικές. Διαπιστώσαμε ότι το 10 με 16% ήταν γυναίκες και ακόμα και αυτές που συμμετείχαν σε πολιτικές αποστολές ε, εκεί ήταν το 7 με 13% γυναίκες. Ε, αυτός είναι ο κόσμο του σήμερα και όχι το 411 π.Χ. Ε, και οι κυβερνήσει των κρατών μελών ε, είναι υπεύθυνε να στήσουν από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης να συγγνώμη, της, ε, του, Ευρωπαϊκού, του, Συμβουλίου, της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αυξήσει τον αριθμό ε, των γυναικών στις συνενευτικές διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρουν ευθύνη για τη διασφάλιση προϋπολογισμού και πόρων ώστε να υπάρξει συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία με την οργάνωση 1325. Ε, στην έκθεσή μα, συζητάμε διάφορα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να τα λάβετε αυτά υπόψη στις μελλοντικέ σα εργασίες. Να εξεταστεί ε, η ε, διαδικασία πρόσληψης υπό το φως των φυλατικών διακρίσεων, να εξεταστούν οι σχετικέ στατιστικέ, να δημιουργηθεί μια κεντρική μονάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευθύνη την συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές αποστολέ, να τεθούν στόχοι όσον αφορά την κατανομή των φύλων, ε, να υπάρχει εκπαίδευση σχετικά με ε, την ισότητα των φύλων ε, και να διορίζονται και άντρες και γυναίκες. Σε σειράξει όλο τον κόσμο από τα Βαλκάνια στην Ρουάντα, από το Αφγανιστάν μέχρι το Ιράκ οι γυναίκες βιάζονται, καταπιέζονται και χρησιμοποιούνται ως σκλάβες και δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες επίλυση διαφορών ε, στις ε, διαμεσολαβήσεις ε, και στις διαπραγματεύσεις ειρήνης. Ένα διεθνές δικαστήριο που θεωρεί την σεξουαλική βία ε, έγκλημα πολέμου όπως ε, είναι και οι βασανισμοί. Ε, αυτό είναι απαραίτητο. Έχουμε σήμερα ένα τέτοιο δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά λυπάμαι που δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν. Το αίτημα να σταματήσει η σεξουαλική βία ε, αναφέρεται σαφώς ε, στο ψήφισμα 1325, άρθρο 10 και 11. Το 2008 το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΟΙΕ υιοθέτησε με ένα συγκεκριμένο ψήφισμα για τον βιασμό και την σεξουαλική κακοποίηση σε ένοπλες σειράξεις. καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί ε, είχαμε τελικά τον, το ψήφισμα 1820 ε, ε, διότι βάζει τέλος στην ατιμορρησία των ε, δραστών. Και ε, πέρσι τον Δεκέμβριο υιοθετήθηκε το ψήφισμα 1960, το οποίο παραδέχεται ότι η σεξουαλική βία είναι σοβαρό έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και κατά του διεθνού δικαίου και ω εκ τούτου θεωρείται έγκλημα πολέμου. Και αυτό ήταν σημαντικό βήμα πρόοδου, διότι ήδη φέτο τον Ιανουάριο, μετά από τον βιασμό 60 γυναικών στο Φίζι, στο Ανατολικό Κονγκό, συλλήφθησαν και καταδικάστηκαν 11 ε, ύποπτοι από το, ε, την άμυνα του Κονγκό. Ε, χρειάζονται περισσότερες ε, γυναίκες επόπτες ε, στην καταπολέμηση τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια ανώπλων σειρώξεων και θα πρέπει να αναλυφθούν συγκεκριμένες δράσεις ώστε να συμμετέχουν οι γυναίκε στι ειρηνευτικέ διαδικασίε. Θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 40% οι γυναίκες στις διαμεσολαβήσει, στις ειρηνευτικέ αποστελές και στην επίλυση διαφορών και στις δραστηριότητε επιβολής τη ειρήνη. Περισσότερε γυναίκε θα πρέπει να συμμετέχουν στη διπλωματία ε, και θα πρέπει να ε, υπάρχει ε, παρακολούθηση των πόσων γυναικών θα πρέπει να υπάρχει μητρό εξειδικευμένων γυναικών και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν οι γυναίκες να συμμετέχουν σε αυξανόμενο βαθμό σε όλα τα επίπεδα ε, λήψης αποφάσεων, ε, την ε, πρόληψη, την επίλυση διαφορών και σε όλη την ειρηνευτική διαδικασία. Το άρθρο 18 του ψηφίσματος 1325 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν όσον αφορά την ασφάλεια και την ειρήνη. Η συμμετοχή των γυναικών είναι προϋπόθεση για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και να θυμόμαστε ότι τα ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Αθνών. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να, εφαρμόζουν, να εφαρμόσουν το ψήφισμα 1325 ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, μετά από πάνω από 10 χρόνια έχουμε δει λίγες ε, συγκεκριμένες προτάσεις ε, για να, ε, ώστε τα λόγια να γίνουν πράξεις. Μέχρι τώρα μόνο 27 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν καθιερώσει εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325. Αυτή είναι πολύ μικρή επιτυχία. Μια, η δική μου χώρα, η Σουηδία, ήταν μια από τις πρώτες χώρες. Ωστόσο, μόλις το 2006, 6 χρόνια μετά δηλαδή, το εφάρμοσε αυτό το σχέδιο δράση. Τη της Φιλανδίας είναι μάλλον το καλύτερο εφόσον εφαρμοστεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι ε, τόλμησαν οι Φιλανδοί να θέσουν το στόχο ε, συμμετοχής γυναικών κατά 50% και θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε χρόνο. Κάθε υπουργό ε, θα πρέπει να λογοδοτεί σχετικά με το τι έχει κάνει για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό. Τα σχέδια δράσης όμως δεν αρκούν. Και σίγουρα όχι αν τα αποτελέσματα δεν είναι μετρήσιμα. Έχουμε αρκετέ πολιτικέ και γενικέ κατευθυντήριε ε, γραμμέ. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι συγκεκριμένε δράσει σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρέπει να ενεργήσουμε δηλαδή. Η Μάρκο Βάλστρομ ε, δήλωσε ότι το θέμα του βιασμού γυναικών ε, δεν είναι θέμα αποκλειστικά της Αφρικής, ε, είναι κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο και έχει 7 χώρες ε, στο θεματολόγιο της και έχει 5 θέματα. Να μην υπάρχει ατιμορρησία. Δεύτερον, να δοθεί η ισχύ στις γυναίκες. Θα πρέπει και οι γυναίκες να αποφασίζουν. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική ευθύνη. Τέταρτον, θα πρέπει να ε, υπάρξει κατανόηση του συστήματο ε, τη βία κατά των γυναικών. Και πέμπτον, να ε, υπάρχει συντονισμό των εργασιών των Ηνωμένων Εθνών. Το φθινόπωρο του 2010 στη Σουηδία ε, μαζέψαμε πάνω από 160 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν την κοινωνία των πολιτών, ε, ε, τη κυβέρνηση, ανθρώπους που διαμορφώνουν πολιτική, ερευνητές και δημοσιογράφους από 20 χώρες του κόσμου σε μια διεθνή διάσκεψη για να γιορτάσουμε την 10η επέτειο του, ε, του ψηφίσματος 1325. Ο στόχος ήταν να εξεταστούν ε, οι καλές και κακές πρακτικές ε, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν κάποια εργαλεία για την εφαρμογή του ψηφίσματος στην πράξη. Και ως αποτέλεσμα των πολύ χρήσιμων συζητήσεων Διαβιβάσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ και στον Γενικό Γραμματέα της ε, τι βασικές συστάσεις. Και είναι για το, τα Ηνωμένα Έθνη η εξή ε, να υπάρξει η ιδιαίτερη ε, ε, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλεία για την συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία και στη λήψη αποφάσεων. Τουλάχιστον 40% γυναίκες συμμετέχουν σε όλε τι ειρηνευτικέ διαδικασίε και ιδιαίτερα στι ε, ομάδες ε, διαπραγματεύσεων ε, να υπάρχουν ποσοστώσεις ώστε να υπάρχουν εξειδικευμένε γυναίκε σε ηγετικέ θέσει στον ΟΗΕ να απαιτείται κάθε χρόνο λογοδοσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1425, να υπάρξουν οικονομικοί πόροι για ε, να στηριχθεί το ψήφισμα 1325. προτείναμε όμως και στα κράτη-μέλη, καλέσαμε όμω και τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τι γυναίκε σε όλα τα επίπεδα λήψη αποφάσεων ε, για την ειρήνη και την ασφάλεια, τουλάχιστον 40% να είναι των γυναικών, να υιοθετηθούν εθνικά σχέδια δράση με μετρήσιμού στόχου, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σαφούς, σαφή, σαφή χρονοδιαγράμματα, ε, αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθηση και συγκεκριμένο προπολογισμό κάθε χώρα θα πρέπει να ορίσει μία πρέσβη για το ψήφισμα 1325 και να υπάρχουν περισσότεροι οικονομικοί πόροι για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ε, λοιπόν εναλλακτικέ λύσεις ε, στο, στον πόλεμο και στη βία, διότι ο πόλεμος ε, σχεδιάζεται, ετοιμάζεται και εκτελείται από ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο πόλεμος και η βία μπορεί να σταματήσει, να ανεχαιριστεί και από, επίσης από ανθρώπους, από γυναίκες και άντρε, από τον αγώνα τη Λυσιστράτη, 400 χρόνια π.Χ. μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια βασική κατεύθυνση. Μην ανακατεύεστε ή ε, όπως ε, είπε ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στο Κοινοβούλιο όταν εκ μέρους της Επιτροπής αυτής έπρεπε να υποβάλω έκθεση για τις γυναίκες και τις σειράξεις μας είπαν ότι εσείς οι γυναίκες δεν πρέπει να ασχολείστε με τέτοια πράγματα δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς οι άντρες για σας παλεύουμε οι γυναίκες όμως πρέπει να ασχοληθούν με τέτοια θέματα και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν ε, και ε, να απαιτήσουν να λαμβάνονται υπόψη και οι δικές μας εμπειρίες. Αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε ε, βιώσιμη ειρήνη, μακροπρόθεσμη ειρήνη. Η ειρήνη είναι πολύ βαριά για να την φέρει μόνο ένας φορέας, μία κυβέρνηση ή ένα από τα δύο φύλλα. Το μισό του παραδείσου το στηρίζουν οι γυναίκες. Ε, η ειρήνη στη γη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ε, επιτραπεί στις γυναίκες να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μάιμπριτ. Είναι σημαντικό αυτό που τόνισε στο τέλος, ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις ε, στον πόλεμο και στη βία. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πω ότι συμφωνούμε ότι οι γυναίκες ε, πρέπει να ανακατεύονται στα θέματα αυτά. Θέλουμε να συμμετέχουμε, έχουμε εμπειρίες ε, που είναι απαραίτητες για να αποφευθούν οι καταστάσεις αυτές. Επίσης χαίρομαι Χαίρομαι πάρα πολύ με τη δουλειά που ε, έχεις ε, κάνει ε, ως, και που αφορά το ψήφισμα 1325. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Ευχαριστώ πολύ Μάιμπριτ, λοιπόν. Στο πρόγραμμα τώρα λέει ότι θα δώσω το λόγο σε δύο ε, μέλη της Επιτροπής μας ε, που είναι σκιώδεις εισηγητές ε, στην έκθεση αυτή πρωτοβουλίας. Πρώτα να δώσω λοιπόν το λόγο στον Ραούλ Ρομέβα που εκπροσωπεί τους Πρασίνους εδώ στο Κοινοβούλιο. Από πέντε λεπτά έχουν οι Ευρωβουλευτές. Έχεις λοιπόν το λόγο, παρακαλώ. Thank you so much. Actually... Ευχαριστώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα αυτό. Στην προηγούμενη μου ζωή συμμετείχα σε πολλές ε, ομάδες του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση σειράξεων από στη Βοσνία. Και εστερνίζομαι πολλά από τα αισθήματα που εκφράσατε μέχρι τώρα και τις απογοητεύσεις. Γιατί τις βίωσα και εγώ προσωπικά όλες αυτές τις απογοητεύσεις. Έχω μερικά γενικά σχόλια και μία ερώτηση. Πριν από πολύ καιρό είχα ακούσει ένα γνωστό ερευνητή για θέματα ειρήνης στον κόσμο που εξηγούσε μια ιστορία για τους Βίκινγκς. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία, θα με διαψεύσετε. Πάντως ήταν καλά τεκμηριωμένη. Μας είπε την ερώτηση, το θέμα, μας είπε ότι διαρωτώνταν γιατί κατά παράδοση οι πολιτισμοί όπως των Βίκινγκς μετατράπηκαν σε κοινωνίε διατήρηση τη ειρήνη. Και υπήρχε ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί τέτοιε αιμοβόρε φυλέ τελικά μετατράπηκαν σε τέτοιε κοινωνίε. Μα ήταν λογικό γιατί όταν ε, οι άνδρε πολεμούσαν, οι <laughs> γυναίκε κάθονταν στι αιστείε του και προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ειρήνη και διαπαιδαγωγούσαν αυτό το φιλιρινικό πνεύμα τα παιδιά του. Εξού και η μετατροπή των κοινωνιών σε πιο φιλιρινικέ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία. Πάντως, ε, φαίνεται καλά τεκμηριωμένη. Και όπως είπατε και εσείς, ο πόλεμος είναι ένας θεσμός, ε, επινοήθηκε, δημιουργήθηκε και εκτελέστηκε από ανθρώπινα όντα. Και αν αυτοί που εκτελούν τους κανόνες ε, και ε, αυτοί που εφαρμόζουν το σύστημα είναι κατά κανόνα άνδρες, βλέπουμε που οδηγούν το σύστημα και ποιε είναι οι συνέπειε. Γιατί είναι γεγονό και μας είμαστε ειλικρινεί και στο παραδεχθούμε ότι ο πόλεμο είναι ένα θεσμό ε, τον οποίο επιβάλλουν οι άνδρες. Ε, οι άνδρες ηγούνται αυτού του θεσμού γιατί αυτοί έχουν τα ενία τη εξουσία σε όλα τα μέρη του κόσμου. σω είχαμε διαφορετική κατάσταση αν τα ενία τη εξουσία τα είχαν οι γυναίκε. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση που υποβάλλατε και οι δύο ότι μία από τις βασικές προσεγγίσεις, ένα από τα βασικά βήματα που έχουμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε την παρουσία των γυναικών σε ηγετικό επίπεδο, σε από το τοπικό επίπεδο μέχρι το διεθνές. Παρουσία των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις, σε ηθήνουσες θέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε προκειμένου να επιφέρουμε κάποια αλλαγή. Μία δεύτερη παρατήρηση και δεύτερη ιδέα που θα ήθελα να εκθέσω είναι ότι συμφωνώ ότι πολύ συχνά βλέπουμε τις γυναίκες στον πόλεμο ως θύματα. Αναφερθήκατε στην έννοια του επιζώντα, ότι οι γυναίκες προτιμούν να θεωρούνται ως ε, επιζώντες παρά ως θύματα. Αυτό είναι μια, δείχνει μια αλλαγή στην προσέγγιση. Κάτι άλλο όμως πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος των γυναικών ως ε, διαμεσολαβητών υπέρ της ειρήνης και φορέων για τη διαφύλαξη ειρήνη. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και νομίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να διατρανώσουμε. Ήμουν ε, και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία μέλο τη Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα και συμμετείχα στην Επιτροπή των Γυναικών ταυτόχρονα και συμμερίζομαι αυτή την απογοήτευση, αυτή τη ματέωση που αισθανόμαστε, επειδή αυτά τα θέματα τα ε, εξετάζουμε μόνο εμείς και η Υποπιτροπή ε, Ασφάλειας και Άμυνας ασχολείται με υποτίθεται πιο σοβαρά θέματα, θέματα άμυνας, ε, οπλισμών, αφοπλισμού. Και για τα θέματα της κατάστασης των γυναικών στη σειράξη μόνο εμάς απασχολούν. Αυτό το θέμα του ρόλου των γυναικών ε, στις σειράξεις, είτε ως θύματα είτε ως ε, φορέο της ειρήνης, δεν κρίθηκε αρκετά σημαντικό ώστε να απασχολήσει τη ΣΕΔΕ, την Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα και παραπέφθηκε σε εμά, την Επιτροπή Γυναικών. Και αυτό και σωστά είπε η κυρία Νικολάη, ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια οριζόντια επιτροπή, μια, μια οριζόντια συζήτηση υπερ άνω των διαφόρων επιτροπών και των διαχωρισμών. Ήμουν στη Βοσνία σε μια περίπτωση που έπρεπε να κατασκευαστεί μια γέφυρα για τον τοπικό πληθυσμό. Και όταν οι μηχανικοί σχεδίασαν τη γέφυρα, ε, ήταν δυνατή διέλευση της γέφυρας μόνο οδικός, μόνο με αυτοκίνητο. Κάποιος ρώτησε λοιπόν, θεωρείτε ότι η προσέγγιση αυτή δείχνει μία μεροληψία υπέρ ενός φίλου. Γιατί, σκεφτήκαμε, για γέφυρα μιλάμε, ένας πολιτικός μηχανισμός, γιατί να σκέφτεται το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Το θέμα είναι ποιο οδηγεί όμω στην περιοχή αυτή τη Βοσνία. Οδηγούν και οι γυναίκε ή μόνο οδηγούν οι άνδρε. Κυρίω οδηγούν οι άνδρε. Οπότε υπάρχει στη γέφυρα αυτή η μονο οδηγουν οι άντρε. κυριω οδηγουν οι άντρε. οποτε υπαρχει στη γεφυρα αυτη η δυνατοτητα να περάσει κανεί πεζό. Όχι, μόνο αυτοκίνητα μπορούν να περάσουν τη γέφυρα. Δεν, προβλέπεται χώρο για να τη διέρθει ε, πεζό. Άρα Μόνο αυτοί που οδηγούν, μόνο αυτοί που έχουν αυτοκίνητο μπορούν να περάσουν τη γέφυρα. Η ερώτηση είναι, φαίνεται απλή, αλλά κάποιος θα πρέπει να προβληματιστεί. Και νομίζω ότι κάποιος ηθήνων που θα λάβει μια απόφαση θα πρέπει να υιοθετήσει αυτή την διαφορετική προσέγγιση. Γιατί μερικές φορές ακόμη και για τόσο απλά θέματα που φαίνονται μηχανικά ε, υπησέρχεται το ζήτημα των δύο φύλων. Και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια οριζόντια συζήτηση μεταξύ όλων των επιτροπών και όχι μεμονωμένη μια συγκεκριμένη επιτροπή. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η έκθεση θα πρέπει να είναι ε, συνοπτική, φιλόδοξη αλλά ταυτόχρονα και εφικτή και να αποφύγουμε σφάλματα του παρελθόντος. Δηλαδή να λέμε πολλά ωραία λόγια αλλά ανέφικτα και αδύνατον να εφαρμοστούν στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέβα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιανακουδάκη που είναι μέλος ε, της ομάδας ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Παρακαλώ κυρία Γιανακουδάκη. Um, Ευχαριστώ. Όταν διάβασα για πρώτη φορά το θέμα, μπερδεύτηκα και πραγματικά δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Γιατί πήρα το θέμα κατά γράμμα, δηλαδή η κατάσταση των γυναικών στις σειράξεις. Αναφέρθηκε ο πόλεμος και η συγγήτρια είχε δίκιο ότι υπάρχουν πολλά είδη πολέμου. Υπάρχουν και πόλεμοι που γίνονται σώμα με σώμα, αλλά υπάρχουν και διάφορα είδη πολέμου. Δεν υπάρχει μόνο η σωματική, η πτυχή. Και ε, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι είμαι ειρηνίστρια και αυτό που θα πω το λέω με βαριά καρδιά. Πολλές φορές δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να πολεμήσει κανείς και υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις που δεν υπάρχουν άλλες ε, διέξοδοι, άλλες αναλλακτικές λύσεις. Θυμάστε τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Δεν μας αρέσει ο πόλεμος, αλλά μερικές φορές δεν έχουμε άλλη λύση. Μερικές φορές όμως υπάρχει επιλογή για παράδειγμα το Ιράκ, αλλά αυτή είναι πολύ δική μου προσωπική άποψη. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε τον πόλεμο και υπό τη σκοπιά του στόχου του λόγου για τον οποίο έγινε. Μπορεί να γίνει για τη δημοκρατία, για την ασφάλεια, για τους άνδρες και τις γυναίκες. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την ανάλυση σας για τα θύματα, τους επιζώντες, ε, την ανάγκη των γυναικών να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική διαδικασία και πολλές φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πολλές γυναίκες σε τέτοιε διαπραγματευτικές ομάδες και χαίρομαι για το σχόλιο σα να συμμετέχουν οι γυναίκες σε επιχειρήσεις διατήρηση ειρήνη. Εμεί το έχουμε αυτό ευτυχώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης ε, και η πολιτιστική σκοπιά ε, επηρεάζει μερικέ φορέ την αντιμετώπιση των γυναικών. Τώρα, αυτά την πλευρά, την, τον, από την πλευρά των πολιτών, το θέμα της πολιτικής προστασίας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να περιληφθεί στην έκθεση είναι η κατάσταση των γυναικών στις σειράξεις, αλλά και η θέση τους στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν θα περιληφθεί και αυτό το θέμα, γιατί εκεί είναι που αντιμετωπίζω ένα ηθικό δίλημα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην ισότητα των δύο φύλων και πιστεύω ότι αν συμμετέχουμε και στο στρατό θα πρέπει να βρισκόμαστε και εκεί επίσης όρις. Βέβαια, από σωματική άποψη είμαστε λίγο πιο αδύναμες, αλλά αν κανείς ε, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή δεν θα πει σφαίρα συγγνώμη, δεν θα σε χτυπήσω σένα επειδή είσαστε το ασθενέ φίλο. Αν κάποιος πάει να πολεμήσει θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό και χαλκέντερος. Μερικές φορές ε, οι γυναίκες αποκλείονται από τις ένοπλες δυνάμεις, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης ε, αποκλείονται μερικές φορές από την πρώτη γραμμή, δηλαδή από την, ε, το να βρίσκονται σε σώμα με σώμα επαφή με τον εχθρό και να μπορεί να τον σκοτώσει. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι, έχουν πιο ισχυρή προσωπικότητα μερικές φορές από τους άνδρες και αν χρειαστεί να κάνουν κάτι θα το κάνουν και αυτές. Πιστεύω ότι και εκεί χρειάζεται μια ισοτιμία. Υπάρχει λοιπόν η σωματική πλευρά, όπως σας είπα, γιατί εκεί είδαμε ότι 1% των γυναικών πληρούν τα σωματικά προσόντα, αλλά ε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει τα σωματικά προσόντα να επιτελέσει τα ίδια ε, το ίδιο έργο με τους άνδρες στο στρατό. Πιστεύετε ότι εκεί θα πρέπει να έχουμε εξαιρέσει, εγώ είμαι κατά των εξαιρέσεων. Έχουμε πολλές γυναίκες, 1.600 ε, γυναίκες έχουμε στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή, πολλές γυναίκες ένοπλες δυνάμεις και από την άποψη αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει το έχει το προβάδισμα εδώ σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών στις σειράξεις. Βέβαια είναι δύσκολο συναισθηματικά πολλές φορές για τις γυναίκες η συμμετοχή Παρόλο που υπάρχουν και ευαίσθητοι άνδρε, δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνδρε είναι ανέστητοι. Αλλά θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Ίσως δεν είναι όλοι τόσο ευαίσθητοι. Θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή. Αλλά θέλω ισότητα για τι γυναίκε, θέλω να αντιμετωπίζονται ισότιμα ακόμη και όταν βρίσκονται στο πεδίο τη μάχη, Γιατί μόνο τότε θα έχουμε ισότητα και στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με του άνδρε. Ευχαριστώ. Yes, but But Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιανακουδάκη. Θα ακούσουμε τώρα τις παρατηρήσεις ε, της εκπροσώπου της ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Καταρίνα Βάλε Κρούντιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ μόλις συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα και εγώ να μιλήσει σουηδικά. Είμαστε στην ε, εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, στα τμήματα διαχείρισης κρίσεως και δυστυχώς ε, ή ευτυχώς η καθομιλουμένη εκεί είναι η αγγλική γλώσσα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε κάποια θέματα τα οποία ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Καταρχάς όσον αφορά τη σημασία του να λαμβάνουμε υπόψη ε, τα θέματα φύλου και γενικώ ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των προτέρων ε, στα θέματα της κοινή εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, στις αποστολές και στις επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξέλιξη των αποστολών και των επιχειρήσεων. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ε, και από όσου χαράσουν πολιτική αλλά και όσου εφαρμόζουν ε, την, ε, το ψήφισμα 1325 και όλα τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ότι ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου, όπως επίσης και στην κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας, διότι αυτά επαρκούν όχι μόνο για τη διαχείριση των κρίσεων, αλλά και για ε, ε, επιτυχή πρόληψη. Η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διάθεση του φύλου είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε αποστολέ όπου υπάρχει και παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη. Ε, μπορεί να διαδραματίσουν και κάποιο ρόλο στις αποστολές ε, για την πρόληψη. Οι αποστολές ε, γίνονται σε περιοχές όπου οι ειρηνευτικές διαδικασίες ενδιαφέρονται και για την κινητοποίηση και για τα παιδιά και ε, υπάρχουν και κάποια θέματα μεταβατικής δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο στόχος μιας κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από πλευράς ασφαλείας είτε από πολιτικούς σκοπούς, είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού και να υπάρχει, να διασφαλίσει ότι υπάρχει ειρήνη. Και επομένω η διάσταση του φύλου είναι σημαντική και όταν διαβιβάζουμε βασικά μηνύματα στον τοπικό πληθυσμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη και να γίνει αποδεκτή η ευρωπαϊκή αποστολή, η ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να επισημάνουμε και ότι οι πολιτικές του φύλου θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Και εδώ επανερχόμαστε και στο θέμα των θυμάτων και το να μην επικεντρωνόμαστε στο πώς θα θυματοποιηθεί κάποιος, αλλά πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να κάνουμε αυτό που έχουμε πάει να κάνουμε. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε απάντηση από στρατιωτικής πλευράς ε, και ήταν ιδιαίτερα δεκτική για τα θέματα του φίλου ως ε, τμήμα της προσέγγισης τους ε, που θα πρέπει να βασίζεται και στα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τις αποστολές και τις επιχειρήσεις, τα έγγραφα κατά την προετοιμασία των διαφόρων αποστολών και επιχειρήσεων ασχολούνται και με θέματα φύλου και με ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού με διάφορους τρόπους. Ε, κατά κανόνα τα διάφορα έγγραφα, τα επιχειρησιακά σχέδια και τα άλλα βασικά έγγραφα αναφέρονται στις υπεφωνημένες σχετικές ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως ε, Καταρχήν, δεχόμαστε τα θέματα αυτά. Από εκεί και πέρα στην πρακτική εφαρμογή υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις. Σε γενικές γραμμές ε, αναφερόμαστε σε αυτά τα έγγραφα σχεδιασμού και στις προσλήψεις, ε, στην κατάρτιση, στις εκθέσεις, τα πειθαρχικά μέτρα, αλλά και στις εξωτερικές προβολές των θεμάτων αυτών. Πώς μπορούμε να μεταφράσουμε την πτυχή του φύλου στις δραστηριότητες που έχουμε επιτόπου και πώς μπορούμε να διοχετεύσουμε καταλληλότερα τις αρχές ε, στις εργασίες που έχουμε με τον τοπικό πληθυσμό. Σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές αποστολές και επιχειρήσεις, οι εντολές των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν και συγκεκριμένες διατάξεις που ασχολούνται με θέματα ε, φύλου και ειρήνης και ασφάλειας ε, πολύ συχνά ως συγκεκριμένο τμήμα τη αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν και κάποια, παρά το γεγονό ότι στα θέματα της εφαρμογής, ε, όπως σα είπα και προηγουμένω είναι αρκετέ ε, οι, προκλήσεις, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές. Για παράδειγμα, υπάρχουν σημεία εστίασης για θέματα φύλου, υπάρχει το θέμα της προαγωγής, της συμμετοχής ε, γυναικών στην ε, συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό και αυτό που έχει σημασία εδώ δεν είναι μόνο ο αριθμός των γυναικών σε στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις, αλλά και πού βρίσκονται στις διάφορες επιχειρήσεις. Είναι πολύ εύκολο να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών, που μπορεί όμως να βρίσκονται σε γραφεία και να μην έρχονται σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, ενώ αν αναφερόμαστε σε περιπολίες ε, και σε άμεση επαφή με το γυναικείο πληθυσμό, εκεί σαφώς ε, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό γυναίκες. Επίσης υπάρχουν και τα παραδείγματα της χρηματοδότησης ε, προγραμμάτων που αφορούν τις γυναίκες, ενημέρωση των τοπικών οργανώσεων για περιστατικά ε, βίας κατά των γυναικών, επαφή ε, με ομάδες ε, γυναικών και ενημέρωση στις αποστολές και επιχειρήσεις και διάλογο με τις διεθνές οργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε σε περισσότερη γυναικεία συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις, υπάρχουν σαφώς προκλήσεις στις συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού ε, της αποστολής ε, και των τοπικών φορέων που σχετίζονται με προβλήματα όπως είναι οι γλωσσικές δεξιότητες ή σε κάποιες περιπτώσεις το αν κάποιος είναι άνδρας ή γυναίκα οι αποστολέ και επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι αντίστοιχε αποστολέ του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Επομένω, θα πρέπει να δώσουμε τη, δέωση, τη δέωσα προσοχή για περισσότερε προσλήψει που θα λαμβάνουν υπόψη και τη διάσταση του φύλου και για να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίε και ισορροπία φύλων στι ίδιε τι αποστολέ, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα είναι και πιο αποτελεσματικέ οι επιχειρήσει, ιδίω όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τι γυναίκε επιτόπου. Και για να επανέλθω σε αυτό, συμφωνώ ότι ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε 50% γυναίκες και 50% άνδρες στις αποστολές και στις επιχειρήσεις. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πώς έχει πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Ε, στην πραγματικότητα έχουμε περισσότερες γυναίκες στις αποστολές και στις ε, επιχειρήσεις ε, από ό,τι έχουμε στα εθνικά μας συστήματα και αυτό θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Η επιμόρφωση βεβαίως είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από πλευράς ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αλλά αυτό είναι πάντα ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς προσπαθούμε όμως να ασχοληθούμε με το ζήτημα στο δυνατό περισσότερο. Τέλος, όπως ε, ρυθμίζεται από τις συμπεφωνημένες έννοιες πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιαδήποτε επιχείρηση και αποστολή περιλαμβάνει πλέον και εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φύλου. Αλλά τα σημεία επαφής ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή γυναικών μπορεί να έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε άλλα καθήκοντα και μπορεί να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικό με αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα αποστολών και επιχειρήσεων όπου υπάρχει προσωπικό πλήρους απασχόληση που ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα θέματα. Θα σταματήσω εδώ και αν υπάρχουν ερωτήσεις με τα χαράς να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας από την, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και έχουμε ώρα για ερωτήσεις. Όποιος θέλει το λόγο, όχι μόνο Ευρωβουλευτής, όποιος έχει απορίες μπορεί να τις θέσει και θα ακούσουμε και τα τελικά σχόλια των προσκεκλημένων μας για να ολοκληρώσουμε την ακρόαση. Κυρία Τόμσον, ευχαριστούμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, γιατί είχα στείλει σχετικές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κατευθυντήρες γραμμές συμπεριφοράς των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ε, διορίζονται σε ε, περιοχές που βρίσκονται σε σειράξεις ε, ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διατήρησης ειρήνης. Γιατί ξέρω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέτοιες ε, κατευθυντήριες γραμμές ό,τι αφορά τις επισκέψεις σε ιερόδουλες και αντιμετώπιση του τοπικού πληθυσμού ανάλογα με το αν κάποιος είναι αποσπασμένος εκεί για βραχή ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, τι συμμετοχή γυναικών υπάρχει σε ό,τι αφορά τις διάφορα, τα διάφορα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν αρκετά, αρκετές γυναίκες που έχουν προσληφθεί εκεί. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν πριν ξαναδώσω το λόγο στις ε, προσκεκλημένες μας. I'm so sorry. Uh, Έχω ένα σχόλιο για τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα που, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ε, υπάρχει κάτι στα γαλλικά που λέγεται «angelisme», ένα είδος ε, ε κατηγορηματικού διαχωρισμού μεταξύ καλού και κακού. Δεν είναι κατά ανάγκη όλοι οι κακοί και αιμοβόροι και αιμοδιψείς και όλες οι γυναίκες ε, το αντίθετο. Είχαμε ε, γυναίκες στη Ρουάντα που χρησιμοποιούσαν τέτοια δρεπάνια και απλώς ε, τέτοιου είδους ε, αρχές πατριαρχικές κοινωνίες είναι δύσκολο να τις εκφράσουν γυναίκες, τις εσωτερικεύουν συνήθως. Και πολλές φορές η φαλοκρατική συμπεριφορά φαίνεται αλλού. Οι γυναίκες πάντως επικοινωνούν σίγουρα πολύ πιο εύκολα. Θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο σας για την παρουσία των γυναικών στο στρατό. Ιστορικά έχουμε τελείω διαφορετικέ εξελίξεις. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Ρώσοι έφεραν τι γυναίκε στο μέτωπο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε ένα τάγμα γυναικών που είχε πραγματικά τρομερές επιδόσεις. Και οι γυναίκε σκότωναν άνδρες στο μέτωπο. Δεν είναι ότι οι Ρωσίδε ήταν ισχυρότερε από τι υπόλοιπε γυναίκε, αλλά ήταν ε, αποφασισμένε και αναγκάστηκαν να το κάνουν. Από ιστορική άποψη, δηλαδή, έχουμε παρουσία των γυναικών και στην πρώτη γραμμή και στο μέτωπο. Υπάρχουν ε, άλλε ερωτήσει, εάν όχι. Να δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μας και να δώσω πρώτα το λόγο στην Καταρίνα Βάλε για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν ε, σχετικά με την ε, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία και κατόπιν θα δώσω το λόγο σε άλλες προσκεκλημένες μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις οδηγίες ή το δεδολογικό κώδικα, κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη είτε στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων διατήρηση ειρήνη. Σε όλε αυτέ τι αποστολέ έχουμε σαφεί οδηγίε για τον τρόπο συμπεριφορά και τη συνεργασία την επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Αλλά έχουμε και κάποιους δείκτες, ορισμένοι αφορούν τέτοιου είδους αποστολές, ή καταγγελίες για παραβίες τέτοιου είδους ε, δεντολογικών κανόνων. Μέχρι στιγμής πάντως με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να σας πω ότι είχαμε ελάχιστα παραδείγματα και ελάχιστες καταγγελίες για παραβίαση τέτοιων κανόνων, τέτοιων δεντολογικών κανόνων από το προσωπικό μας. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες φαίες ζώνες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο ακριβείς είναι αυτές οι Αναφορέ Πάντω σίγουρα υπάρχουν δεντολογικοί κανόνε, οδηγίε και για τι στρατιωτικέ επιχειρήσει και για τι ε, επιχειρήσει διατήρηση ειρήνης. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχή των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία αριθμητικά. σω η Καταλήν στη δική τη παρουσίαση το αναπτύξει περαιτέρω. Πάντω είναι σαφέ ότι σε ορισμένε θέσει, όπω είπαμε και προηγουμένω, δεν έχουμε πολλές, πολλές γυναίκες επικεφαλής ή σε επιτελικές θέσεις. Είναι ελάχιστες για να μην πω καθόλου στις στρατιωτικές κυρίως επιχειρήσεις. Δεν έχουμε γυναίκες ε, στρατηγούς, για παράδειγμα. Αλλά στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έχουμε σε ηθήνωσες θέσεις πολλές γυναίκες. Απλώς στη στρατιωτική πτυχή δεν έχουμε μεγάλη παρουσία γυναικών, ιδιαίτερα στις ε, υψηλότερες θέσεις, στις ψηλόβαθμες θέσεις. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ελίσσα Πετρέν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Έγινε συζήτηση σχετικά με τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τις γυναίκες στους πολέμους. Νομίζω ότι και πάλι Μιλάμε για τους πολέμους που γνωρίζαμε εμείς στο παρελθόν. Φυσικά όλοι μας θέλουμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας όταν ε, απειληθεί από κάποιον άλλον. Αλλά δεν θα έλεγα ότι βλέπουμε πολέμους ε, τέτοιες παραδοσιακής φύσης ε, σήμερα. Κάτι στον Κάφκασο βλέπουμε, αλλά όχι ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι το να στείλουμε γυναίκες στην πρώτη γραμμή μάλλον δεν είναι καν επίκαιρο θέμα και ελπίζω να μην γίνει κιόλα. Είναι αλήθεια ότι και οι γυναίκες δεν είναι πολύ καλοί άνθρωποι όταν δούμε τους, ε, τις που υπήρξαν, ε, δεν ξέρω, με η Μάρκετ Θάτσερ, η Ιντιρα Γκάντι, η Γκόλτα Μέιερ. Φυσικά λοιπόν υπάρχουν σκληρές γυναίκες. Μην νομίζουμε ότι είμαστε άγιες, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι εύκολο να λέμε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αποτελούν συγκεκριμένο ποσοστό, να, υπάρχουν να υπάρχει συγκεκριμένο αριθμός γυναικών σε διάφορες θέσεις. Θα πρέπει όμως και οι γυναίκες να ε, κάνουν αιτήσει για τις θέσεις αυτές και να είναι διατεθειμένες να έρθουν. Έχω μιλήσει τόσες φορές με ε, τον... Ε, ε, με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα αυτό και προσπαθούν να έχουν περισσότερες γυναίκες σε ειρηνευτικές αποστολές. Είναι πολύ δύσκολο όμως αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν γυναίκες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό σύστημα το οποίο να μπορεί να εξετάσει και την πολιτική πλευρά. Πρόκειται για επικίνδυνα μέρη δεν μπορεί κανείς απλά να στείλει μια γυναίκα που μπορεί να έχει μικρά παιδιά κτλ. Θα πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη μα τα θέματα αυτά. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ελκυστικές τις θέσεις αυτές. Και φυσικά είναι θετικό το να υπάρχουν ε, σημεία επαφής. Θα πρέπει όμως να έχουν τέτοια θέση στην ιεραρχία ώστε να μπορεί να πάει στον ειδικό εκπρόσωπο και να πει ότι αυτά που κάνει είναι ανόητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και καλοπληρωμένες θέσεις ψηλά στην ιεραρχία, οι οποίες να έχουν τις δυνατότητες αυτές. Ήταν πολύ θετικό το, το ότι η Μάιμπρη ήταν ανέφερε τα εθνικά σχέδια δράσης. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα πιο σημαντικό από τα έγγραφα που εκπονούνται είναι οι δραστηριότητες για την εκπόνηση του σχεδίου, να συνεργαστούν τα Υπουργεία, να υπάρχει κίνηση σχετικά με τα θέματα. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στα περιφερειακά σχέδια δράσης, τα οποία δημιουργούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ε, πώς ε, η Ρουάντα, το Μπουρούντι ε, και η Δημοκρατία του Κονγκό εκπώνησαν μαζί ένα σχέδιο για το μέλλον. Αυτή είναι πραγματικά η ειρηνευτική διαδικασία. Το ίδιο βλέπουμε και στον ειρηνικό. Και στα Βαλκάνια περιφερειακό λόμπι των γυναικών όπου συμμετέχουν οι δημοκρατίες της πρώην Ιουγκοσλαβία ε, και ε, της Αλβανίας. Ε, υπάρχει και εδώ συνεργασία όπου συμμετέχουν οι γυναίκες. Αυτά λοιπόν είναι θετικά μηνύματα όσον αφορά το βιασμό ως έγκλημα πολέμου. Ακόμα και αν δεν μου αρέσει η σκέψη της εκδίκησης, Ήταν καλό το ότι οι πρώτες υποθέσεις βιασμού στο ε, δικαστήριο για την ε, πρώην Ιουκοσλαβία ε, οδήγησαν σε ποινές άνω των 20 ετών. Αυτό δείχνει ότι λαμβάνονται στα σοβαρά υποθέσεις αυτές. Τώρα υπάρχουν αρκετές υποθέσεις ανοιχτές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. από ό,τι φαίνεται θα έχουμε υποθέσεις ε, σεξουαλικής βίας ε, και από τη Λιβύη. Νομίζω λοιπόν ότι βλέπουμε και θετικά μηνύματα, ωστόσο. Ε, είναι αλήθεια ότι πολύ λίγες γυναίκες συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, αλλά στην Αρούσα έστειλαν ε, αντιπροσωπείες ε, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Φυσικά βρίσκονταν στο περιθώριο, ωστόσο ε, επηρέασαν τις διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε τις δραστηριότητες της κοινωνία των πολιτών στις διαπραγματεύσεις αυτές. Νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν θα είχα συνεχίσει μέχρι την ηλικία μου αν δεν ήμουν αισιόδοξη. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να είμαστε αισιόδοξε ώστε να έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε τις εργασίες αυτές. ως αισιόδοξο άνθρωπος βλέπει κανείς και λύσει για το μέλλον και αυτό είναι ο λόγο για όλες τις προσπάθειες αυτές. Ελίσα Πετρέν, ευχαριστώ πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Μάιμπριτ Θεωρήν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ε, ξεκινήσω από εκεί που ε, έκλεισε την παρέμβασή της ε, η Ελίζαπετ. Η Νότια Αφρική και η Γουατεμάλα ήταν επίσης πολύ καλά παραδείγματα όπου συμμετείχαν οι γυναίκες στην διαδικασία. Και θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Ρόμεβα για τους Βίκινγκ. Η Σουηδία είχε 200 χρόνια ειρήνης ε, ε, τώρα βέβαια έχουμε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν δυστυχώ. Ε, Πάντω δεν νομίζω ότι είναι αληθινή η ιστορία αυτή. Ε, Α ε, κοιτάξουμε την πρόσφατη ιστορία. Στο Ελ Σαλβατόρ ε, συμμετείχαν οι γυναίκες στις διαπραγματεύσεις και είχαν ισχυρή θέση. Ήμουν εκεί. Μετά όμως τέθηκαν στο περιθώριο και έτσι δεν είχαν την παραμικρή ελπίδα. Και αυτό γίνεται πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακόμα και στη Σουηδία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την κινητοποίηση του στρατού, οι γυναίκες άρχισαν να παίρνουν ισχυρέ θέσει στην κοινωνία. Θα πρέπει όμως να είμαστε πιο συνεπείς αν θέλουμε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Για μένα η ισότητα δεν είναι να έχουμε ε, εξίσου πολλές γυναίκες όσο έχουμε άντρες στρατιώτες. Ε, προς Θεού, αυτή δεν είναι η λύση. Η λύση δεν είναι στρατιωτική. Η λύση είναι πολιτική για μένα. Διπλωματία και πολιτική. Ε, εγώ σίγουρα δεν θέλω κάτι τέτοιο. Και σίγουρα έχετε δίκιο, οι γυναίκες δεν είναι καθόλου άγγελοι. Δεν καθόλου άγιες. Η Ελίζαμπετ μας ε, ε, έδωσε αρκετά ονόματα, μπορούμε να σα δώσουμε ακόμα περισσότερα όμως, ονόματα γυναικών επιθετικών. Ωστόσο, κατά διάρκεια της ιστορίας, ε, και νομίζω ότι θα, θα συμφωνήσετε, η εμπειρία μας εδώ και χίλια χρόνια είναι διαφορετικές από αυτές των ανδρών και έπρεπε πάντα να βρούμε άλλους τρόπους ε, επίλυσης των ε, λύσεων, από, ε, επίλυσης των διαφορών από τη χρήση της δύναμής μας. Και ρωτήσατε αν, τι διαφορά θα έχει αν συμμετέχουν γυναίκες ε, στις διαπραγματεύσεις. Ε, σίγουρα θα υπάρχει διαφορά, ε, όχι όμως αν υπάρχει μία ή δύο ή τρεις γυναίκες. Θα πρέπει να υπάρχει κριτική μάζα, η κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε να επιφέρουμε διαφορές. Αλλά ακόμα και στη δική μου χώρα, όπου συμμετέχουν σχεδόν κατά 50% στο κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, και εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Θέλει χρόνο μέχρι οι δικές μας εμπειρίες να αλλάξουν την κατάσταση. Είμαι πεπισμένη όμως ότι αυτό θα συμβεί. Και η Ελίσα ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα με ε, την, ε, τη συμμετοχή ε, γυναικών αστυνομικών και το έχουμε συζητήσει αυτό στη Σουηδία και γνωρίζουν ότι είναι πρόβλημα. Εσείς, αν είστε γυναίκα με μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να λείψετε για μισό ή ένα χρόνο. Μπορείτε να λείψετε για τρεις μήνες να γυρίσετε σπίτι, να ξαναφύγετε μετά. Ε, είναι δηλαδή θέμα του να λύσουμε τα πρακτικά προβλήματα κατά τη συμμετοχή των γυναικών. Ε, δεν είναι μόνο το ότι είναι μητέρε, είναι το ότι ε, ζουν υπό διαφορετικέ συνθήκε από ότι άντρε. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι συνθήκε αυτέ. Ε, και γι' αυτό ε, ακούμε ε, προσεκτικά τους διάφορους σουηδικούς φορείς και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Όχι, δεν είμαστε καθόλου άγιες. Σίγουρα όμως απαιτούμε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά μας, να συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην κοινωνία μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. εάν συμμετέχουν οι γυναίκες στη συζήτηση. Θα σας πω αυτό που είπα στη Σουηδική τηλεο... τηλεόραση όταν συμμετείχε η Σουηδία όταν ε, συμμετείχαν ε, οι γυναίκες στον, συγγνώμη, η Σουηδία στον αγώνα κατά του, του ε, Κατάφη, ε, όλοι είπαν ότι ναι, πρέπει και εμείς να είμαστε όσο καλοί είναι και οι άλλοι. Αλλά ούτε η Νορβηγία συμμετέχει, ούτε η Γερμανία. Ε, Υπήρχαν πολλά πράγματα όπου θα, μπορούσαν, ε, όπου θα μπορούσε η Σουηδία να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών ε, αντί να στείλει 8 αεροπλάνα. Αν λοιπόν υπήρχαν γυναίκες ε, στην διαδικασία λήψη αποφάσεων θα μπορούσαν να πούνε σταματήστε, περιμένετε, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα για τους πολίτες, για τους ανθρώπους στην χώρα αυτή αντί να στείλουμε πολεμικά αεροπλάνα. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα αγένεια ή ευγένεια, είναι θέμα κοινή λογικής, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μάιμπριτ. Ε, και οι δύο προσκεκλημένες μας ε, σχολίασαν ε, τις ιδιαίτερες εμπειρίες των γυναικών και το κατά πόσο οι γυναίκες είναι άγιες ή όχι. Θα ήθελα και εγώ να το σχολιάσω αυτό να πω ότι όλοι εμείς ε, που εργαζόμαστε υπέρ τη ισότητα ε, και που θέλουμε να αυξήσουμε την ε, συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις διαδικασίες, δεν θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άντρες, ότι είναι άγγελοι, ότι είναι άγιε. απαιτούμε όμως να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες με τους άντρες να μπορούμε να συμμετάσχουμε, να συμβάλλουμε με τις εμπειρίες μας, με τις ε, ικανότητές μας. Ε, αυτός είναι ο στόχος της, ε, των προσπαθειών μας για την ισότητα και όσον αφορά το θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα και γενικά όσον αφορά τα θέματα ισότητας. Χρειαζόμαστε τις ικανότητες και των δύο φύλων για να δημιουργήσουμε μια όσο γίνεται καλύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση του πάνελ που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και που ε, συμβάλλει σημαντικά στις ε, εργασίες ε, της Επιτροπής μας. Θα προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ακρόασης και την συζήτηση του πάνελ που έχει θέμα οι συνέπειες των σειράξεων στις γυναίκες. πρώτη προσκεκλημένη μας είναι η Κάρολ Μαν, που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και είναι ειδικευμένη σε θέματα ε, των δύο φύλων ε, και, ε, και στις ενοπλές συγκρούσεις. Καλώς ήρθατε. Σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Είμαι τεχνολογικός ανάπηρη. Αν ξέρει κάποιος πώς λειτουργεί αυτό, θα σας ήμουν ευγνώμων. Sorry. So that's Okay, I'll start Θα ξεκινήσω λοιπόν. Θα σας μιλήσω για τις επιπτώσεις ε, των ένοπλων σειράξεων για τις γυναίκες. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Είναι τιμή μου να, βρίσκετε, να βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για μένα. Είμαι ιστορικός και κοινωνική ανθρωπολόγος που ασχολούμαι με θέματα φύλου και διδάσκω στη Γαλλία. Αλλά έχω και πρακτική πείρα ε, διότι ε, διεύθυνα δύο μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε πόλεμες περιοχές, στη Βοσνία και σε μία περιοχή στο Πακιστάν, ε, στο Αφγανιστάν και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα ξεκινήσω τώρα με την παρουσίασή μου. Θα τη διατρέξω στα γρήγορα, αλλά όποιο ενδιαφέρονται έχω διαθέσιμα και CD, διότι βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να το διαβάσουμε δεν ξέρω πώς μεγαλώνει η διαφάνεια και αν μπορώ να τη μεγαλώσω. Τέλος πάντων, έχω επιπλέον ε, CD για όποιον ενδιαφέρεται για την παρουσίαση λόγοι και ιδεολογίες πίσω από τους ε, πρόσφατους σύγχρονους πολέμους. Βεβαίως ε, κάποια από αυτά τα έχετε ξανακούσει. Οι πόλεμοι διαφέρουν ε, πολύ σήμερα, διότι στο παρελθόν ήταν κατακτητικοί πόλεμοι, επεκτατικοί πόλεμοι για να επεκταθούν αυτοκρατορίες και γιατί η γη είχε τεράστια αξία, όπως και ο πληθυσμός που διέμενε σε αυτή τη γη, γιατί μπορούσαν να ενισχύσουν τους αυτοκρατορικούς στρατούς. Μετά από τη Βοσνία που ε, προσπαθούσε να επινοήσει από πλευράς ε, Σέρβων εθνικιστών ε, τη σύγχρονη Ιουγκοσλαβία, έχουμε διαφορετικές εξαιρέσεις. Ο πόλεμος πλέον θεωρείται ως αδικαιολόγητη κατοχή από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε και να είναι αυτή. Ε, έχουμε και εξελίξει σειράξει Ισραήλ, Παλαιστίνη, ε, Ναγκόρνο, ε, Καραμπάχ, το και Αρμενία. Ε, οι βασικοί λόγοι σήμερα πλέον είναι πολιτική και στρατηγική και κατά την άποψή μου η, κυρίως οικονομική πλέον. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός όρος που μας ενδιαφέρει, οικονομικής φύσεως πόλεμη. Συγγνώμη, έχασα και το βοηθό μου. Κάτι πατήσαμε, δεν δουλεύει πλέον. Okay. Because this is meant... Sorry. I hope I still have my 15 minutes to talk. This is... Ελπίζω να μην έχω κατασπαταλήσει και όλο μου το χρόνο. Θέλω απλώς να πάω στην επόμενη διαφάνεια. This one? It's okay? Yeah, that was meant to be bigger, but anyway. All right. Uh, as I... Λοιπόν, όπως σας έλεγα, οι λόγοι είναι πλέον πολιτικοί και στρατηγικοί και κατά την άποψή μου κυρίως οικονομικοί. Η κατοχή γης σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνο για του ανθρώπου που θέλουν να βρουν θέσεις εργασία και τις υποδομές. Επομένω, είναι πολύ δαπανηρή διαδικασία να σκεφτούμε ένα πόλεμο όπως ε, είχαμε στο παρελθόν. Το να κατασκευάσουμε νοσοκομεία και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις ε, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, αν δεν υπήρχαν μάλιστα ακόμα περισσότερο. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι οικονομικοί οι λόγοι πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει πλούτο χωρίς να κάνει και τις ανάλογες δαπάνες. Καταρχάς θα πρέπει να εξασκήσουμε πολιτική επιρροή για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε συμμάχους. Σύμμαχοι θα γίνουν κάποιοι αν υπάρχει ταύτιση ιδεολογικών απόψεων. Οι μουσουλμάνοι ε, Σούνοι, για παράδειγμα, όπως έγινε στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, ε, δημιουργήθηκαν προβλήματα στη συνέχεια γιατί ε, υπήρξαν προβλήματα με τις Φιλένκες και είχαμε τους Ταλιμπάν. Και η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υποστήριζαν ε, τους Ταλιμπάν και στις χώρες αυτές όπως γνωρίζετε δεν υπήρχαν καθόλου ανθρώπινα δικαιώματα ούτε στην πράξη αλλά ούτε και επί χάρτου. Και επίσης θα υπάρξει και συνεργασία αν είναι ταυτόσιμα τα οικονομικά του συμφέροντα. Ε, παρά το γεγονό ότι μπορεί να έχουν τελείω διαφορετικέ πολιτικέ, όπω γίνεται στι ΗΠΑ και στη Σαουδική ε, Αραβία. Ε, οι δικτατορίες και οι αποδυναμωμένες κυβερνήσεις όπως έχουμε στην Αφρική μας επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν πόροι όπως περιοχέ περιοχές των μεγάλων λιμνών που έχουμε εκμετάλλευση των διαμαντών που, και μάλιστα η εκμετάλλευση αυτή είναι μοναρχική, απολυταρχική και για τις γυναίκες δεν υπάρχει κανένα όφελος. Να προσθέσουμε δε και την εξαγορά των, ε, ε, και την κατάληψη των αγορών. Όλα αυτά κατ' εμέ είναι δημοκρατία ε, με την επίφαση του φιλελευθερισμού και έχουμε και μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι ε, κατά του φίλου από το Hollywood στο Mollywood. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Mollywood είναι η τεράστια βιομηχανία ε, που έχουμε στις περιοχές αυτές. No, no. You must control your language, dear. It's not being in the army. Yeah, okay. Because each time it's different. Yeah, you can, you can press this. Okay, right. So, a few illustrations called. Εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είδατε την προηγούμενη γιατί ήταν πολύ καλή. Τέλος πάντων. Ένα κατάστημα διαμαντιών που έγραφε ο Ιησούς είναι πλούσιος. Ε, αυτό δείχνει πώς η ιδεολογία μας ε, επηρεάζει τις καταστάσεις. Αυτή είναι μια σχολική σάκα Συγγνώμη, αλλά κάθε φορά έχω κι άλλο πρόβλημα. Και αυτή η φρικτή εικόνα είναι από μία ταινία του Μόλιγουτ. Δείτε τι κάνει η βιομηχανία ταινιών της Νιγηρίας. Δείχνει τα πιο ε, άσχημα και σεξιστικά πράγματα στον κόσμο. Ποιε είναι οι συνέπειε λοιπόν για τι κοινωνίε που ζουν σε εμπόλεμη κατάσταση. Καταρχά υπάρχουν συνέπειε για την κοινωνία των πολιτών, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την υγεία και την παιδεία και αυτό φυσικά πλήττει ιδίω τι γυναίκε. Και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένε οικονομικέ προτεραιότητε για του πολέμου, οι πλούσιοι γίνονται πλησιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Πολλό δε μάλλον ε, ε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Η εμπορία αυξάνεται εν γέννη, έχουμε ναρκωτικά, ιερόδουλους, ε, σκλάβες για σεξουαλικούς σκοπούς. Το Αφγανιστάν έχει γίνει η πρώτη χώρα των ναρκωτικών μετά τον πόλεμο. Επομένως, επειδή ακριβώς ε, αυξάνεται όλη αυτή η κατάσταση και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, αυξάνονται και οι προκαταλήψεις λόγω φύλου. Αν πάτε σε οποιαδήποτε πόλεμη περιοχή, θα δείτε τι ε, ε, παιχνίδια εξάγονται σε χώρες αυτές από την Κίνα και στο Αφγανιστάν και να δείτε τι πουλούνται στις αγορές και στα σούπερ μάρκετ της Καμπούλ. Και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα προϊόντα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το ίδιο καταπιεστικό παράδειγμα που είναι πιο πιο σημαντικό από οποιαδήποτε προσπάθεια για ειρήνη. Στη συνέχεια έχουμε τις επιπτώσεις του πολέμου για τις γυναίκες. I want to go back. I do apologize. What's what's happening now? Is it? Okay, right. Oh, that's the thing. Okay, right. But here, no. All right. Women in armed conflict. Okay. You've got... Οι γυναίκε τώρα στι ενοπλέ συγκρούσεις, έχετε το κατάλογο, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Η κατάσταση μπορεί να συνοψιστεί ω αύξηση τη βία σε οποιοδήποτε επίπεδο, και ο βιασμό πλέον θεωρείται κάτι φυσιολογικό. Αυτό συμβαίνει σε κάποιε περιοχέ τη Αφρική που δεν υπάρχουν ορυκτοί πόροι δυστυχώ. Ο, ο λοιπόν ω πολεμικό όπλο συνεχίζει ανεμπόδιστο. Υπάρχει και βιασμό ανδρό, όπω είπαμε σήμερα το απόγευμα, αλλά δεν καταγράφεται. Λε και ο βιασμό για τι γυναίκε είναι κάτι φυσιολογικό. Οι γυναίκε γεννούν σε φρικτές καταστάσεις, η θνησιμότητα κατά τη γέννηση αυξάνεται και το Αφγανιστάν έχει το χειρότερο ρεκόρ παρά το γεγονός ότι έχει τόσο μεγάλη υποστήριξη η χώρα. Και φυσικά η παιδεία θυσιάζεται και για, τα, ε, για όλα τα παιδιά και για τα γόρια και για τα κορίτσια και είναι όλοι θύματα πολέμου. Εδώ έχουμε μαχητές γυναίκες του Ταμούλ. εδώ έχετε την αντίσταση, εδώ είναι μια γυναίκα στο Ιράν. Πρόσφυγες, όπως γνωρίζουμε, οι πρόσφυγες είναι στο 80% τους γυναίκες παγκοσμίως. Εδώ έχουμε την κυρία Σαλίβ που συμμετέχει σε ερευνητικέ διαδικασίες. This is my friend Azra in Bosnia. Αυτή είναι η φίλη μου η Άζρα στη Βοσνία που είναι αντιστασιακή. Όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να σας πω κάποια πράγματα διότι ασχολήθηκε με την ε, ε, κατασκευή ενός σχολείου σε μια πολύ άσχημη περιοχή κοντά στο Σαράγεβο. Να περάσουμε τώρα στις συστάσεις. Πρέπει να ξανασκεφτούμε εντελώς ε, την έννοια της βοήθειας. Είναι αδύνατο να βοηθήσουμε γυναίκες σε ένοπλες ε, περιοχές ε, και να τις απομονώσουμε από τις ιδεολογίες. Θα πρέπει να δούμε Πώ έχουν οι συνθήκε. Εγώ σκέφτομαι κάποια σχολεία που είδα στο Αφγανιστάν. Ε, ε, κατασκευάζονται σχολεία, αλλά δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν βιβλία, δεν υπάρχουν θρανία και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τα παιδιά και δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Η Αμερικανική PRD ε, περιγράφει πολύ ωραία την τελετή των εγγενείων, κόβεται η κορδέλα, μια υπέροχη τελετή και μετά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν και κάποιες λύσεις ε, ε, τύπου cut and paste, ε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα υγειονομική περίθαλψη που προσφέρεται σε κάποιες περιοχές και είναι επιτυχής και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού, αλλά δεν χρησιμοποιείται παρκώς. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν να εφαρμόσουμε μια πιλωτική τεχνική. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όμως με όλη την κοινότητα, με γυναίκες και με τις οικογένειές τους οι πόλεμοι γίνονται σε πατριαρχικές κοινωνίες όπου οι γυναίκες είναι κυρίως η κόρη κάποιου, η μητέρα κάποιου, η γιαγιά κάποιου και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα γυναικείας ε, αλληλεγγύης. Στις ε, μεγάλες λίμνες είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά στο Αφγανιστάν ε, η γυναική αλληλεγγύη είναι απλώς οικογενειακή, σε ποιον ανήκει. Η δυτική έννοια της ε, προσωπικής, εγωιστικής προσωπικής ανάπτυξης, ε, καθώς επίσης και ε, ο φεμινισμός της προηγούμενης γενναίας χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις και αποτυγχάνουν παντελώς, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τις ε, τοπικές συνήθειες. Κανένας δεν έχει κάνει ε, μάθημα ανθρωπολογίας, δεν ξέρει πώς έχει κοινωνία και αυτές οι μέθοδοι που αντιγράφουμε από τη μία και τις εφαρμόζουμε σε μία άλλη περιοχή δεν θα λύσουν μαγικώς τα πράγματα όπως ελπίζουμε. Ορισμένε φορέ μπορεί να είναι πολύ ωραίε ε, τα γένεια νέων σχολείων, ε, δημόσιες σχέσεις, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε την τοπική κοινωνία, πώ λειτουργεί η κοινωνία εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ατιμορρησία, ε, σεξουαλικά εγκλήματα και διαφθορά λόγω του πολέμου επίσης. Αυτό σας έλεγα προηγουμένως, αυτό πωλείται στα καταστήματα ε, για στιγμιαία παρθενία. Βλέπετε επίσης παιχνίδια τα οποία ε, είδαμε σε κάποια φωτογραφία στο Αφγανιστάν, παιχνίδια γονιμότητας. Έχουμε κάποιες ακόμα φωτογραφίες. Πρακτικά μέτρα τώρα. Επειδή ακριβώς είναι τόσο απελπισμένες οι συνθήκες, ε, υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καλό ε, σημαντικό είναι να υπάρχει γνώση και θετική στάση για τη ζωή. Και εδώ ε, μας ενδιαφέρει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα σχολεία δεν επαρκούν ε, και η σχολική παιδεία δεν είναι επαρκής. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν δεν υπήρχαν καθόλου σχολεία στο παρελθόν, όπως και σε κάποιες περιοχές της Αφρικής. Δεν υπάρχει λοιπόν και ε, υλικό υποστήριξη, υποστηρικτικό υλικό που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει μια γενναία μέχρι να αρχίσουν να διαβάζουν κάποιοι. Στην καλύτερη περίπτωση μαθαίνουν απλώς να γράφουν το όνομά τους. Θα πρέπει να διερευνήσουμε και άλλα πράγματα ε, τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί ποτέ. Ε, συγγνώμη, αλλά οι διαφάνειες έχουν αποτύχει παταγωδός. η δασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αφηρημένη και άχρηστη αν δεν υποστηρίζεται και από πρόοδο, μετρήσιμη πρόοδο. Η βελτίωση της ε, ε μητρότητας και της φροντίδας των παιδιών όπως και της αναπορεγωγικής υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι αποτυχημένη αν δεν πάει ε, ε, μέσα από τους κατάλληλους διάβλους. Είτε αυτά είναι νοσοκομεία είτε οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται λοιπόν μια προληπτική προσέγγιση για την υγεία. Αυτό είναι ζωτική σημασία και θα πρέπει να υπάρχει και σε έντυπο υλικό. Εγώ κάνω εκστρατεία γι' αυτό ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν θέλουμε να συζητήσουμε θέματα υγείας και παιδείας ε, μέσω άλλου υλικού που δεν είναι ε, αποτυπωμένο σε χαρτί, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δημιουργήσουμε μια τέτοια παιδεία εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντική, για να ξέρουμε και τι δικαιώματα έχουμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά οι διαφάνειες δεν είχα κανένα αποτέλεσμα. Και τέλος έχουμε κάποια μικρά προληπτικά μέτρα Μέσω του ΦΕΜΙΝΤ έκανα πειραματικά μικρά προγράμματα, αλλά ήθελα απλώς να σας αναφέρω κάποια επιγραμματικά. Για παράδειγμα, το να υπάρχουν ε, αποχωρητήρια για κορίτσια σε σχολεία στα οποία υπάρχει ε, μεγάλο, με πολλά περιστατικά βιασμού μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μαθήματα αυτοάμυνας ε, στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα να πολεμήσουμε όταν είμαστε ενάντια σε πέντε ανθρώπους με αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να φέρουν αποτελέσματα και μπορεί να ε, δημιουργηθεί και καλύτερη ε, πρακτική εάν συμπεριληφθούν στο σχολικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να πάψει να υπάρχει το μοντέλο της ε, ανδρικής κυριαρχίας και να ξεχάσουμε και αυτή τη στρατιωτική κουλτούρα γυναίκες οι οποίες ε, δίνουν ένα συνεχή αγώνα για να συνεχίσει να υπάρχει ζωή. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίοι το μέλλον της κοινωνίας και το κάνουν αυτό σε καθημερινή βάση και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τον πόλεμο. Είναι οι γυναίκες που διατηρούν το νήμα και εξελίσσουν το μέλλον, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αναγνωρίζεται ποτέ. Ε, οι καθημερινές ηρωίδες ε, εξαφανίζονται αμέσως. Ε, μπορούμε να κάνουμε έρευνα για τις γυναίκες στη Βοσνία σήμερα, γιατί μετά από κάποιο πόλεμο ε, η ε, ο κόσμος θέλει να ξεχάσει, θέλει να ξεχάσουν το γεγονός ότι πέρασαν τα χειρότερα. Ε, οι στρατηγοί και οι άνδρες ήρωες ακούγονται παντού. Τι γίνεται όμως με τη γυναικεία φωνή. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω, να δούμε αν μπορούμε να το δούμε, εδώ έχουμε ενημέρωση για την υγεία, παιδεία για την υγεία για γυναίκες υπαίθρου που δεν μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν, που είναι αναλφάβητες αλλά πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα. Όσον αφορά ε, τα θέματα του πολέμου, θα έπρεπε να διδάσκεται το θέμα του φύλου και του πολέμου σε όλο τον κόσμο. Να καταγράφονται οι εμπειρίε των γυναικών σε εμπόλεμε περιοχέ και τα στοιχεία να περνούν σε μέσα μαζική ενημέρωση, να καταγραφούν σε βιβλία ιστορία, σε ιστότοπου, στο ραδιόφωνο. Πρέπει να αλλάξει αυτό το παράδειγμα τη ανδρική κυριαρχία. Σα έδειξα αυτή την επονίδιστη εικόνα του Νόλιγουτ. Ε, υπάρχουν σεξιστικά παραδείγματα και θα μπορούσε κάλλιστα να σέβεται κάποιος τις γυναίκες μέσω κατάλληλης παιδείας, αλλά θα πρέπει κάπου να καταγράφετε το τι κάνουν οι γυναίκες και ίσως αυτό θα ενδιέφερε την Επιτροπή σας. Ε, ούτως ή άλλως αποτελεί ένα πρώτο σταθμό για να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία που υπάρχει για τον πόλεμο. Ζητώ συγγνώμη για τις διαφάνειες. Ε, όποιος ενδιαφέρεται όμως, όπως σας είπα, υπάρχουν και σε CD. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά για την ομιλία σας αυτή. Ε, ευχαριστούμε που το διαθέτετε και σε CD, ώστε οι ευρωβουλευτές ε, να μπορούν να το πάρουν. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την επόμενη προσκεκλημένη μας, που είναι η Αν Κατρίν Ριμπνίτσκι που έχει εργαστεί ως σύμβουλος ε, καθώς ε, και στο στρατό. Θα χαιρόμαστε που σε καλωσορίζουμε. Σου δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Χρειάστηκε να αλλάξουμε θέσεις λόγω του υπολογιστή. Και αυτό μας εκπλήσει με όλη αυτή την θαυμάσια τεχνολογία που έχετε εδώ σήμερα. Είμαι 37 ετών Δανική καταγωγή. Πρώτη φορά που μιλάω στο Κοινοβούλιο, χαίρομαι που είμαι εδώ. Πέρασα πολύ καιρό στο Αφγανιστάν, Όπω βλέπετε από αυτή τη φωτογραφία. Πέρασα αρκετά χρόνια στο στρατό, μια δεκαετία για την ακρίβεια. Υπηρέτησα στο Χέλμαντ δύο φορέ στο νότιο Αφγανιστάν, αρχικά ως λοχαγός, εξού και η φωτογραφία, και τη δεύτερη φορά εργάστηκα στο Χέλμαντ ως σύμβουλος άμαχο πληθυσμού στο PRT στο Χέλμαντ και μάλιστα διεξήγαγα πάνω από 200 περιπολίες, ε, είτε πεζή, είτε με Με Είχα πάρα πολλές συναντήσεις και ίσως η δική μου εμπειρία από το Αφγανιστάν είναι κάπως διαφορετική από τη δική σας. Βέβαια, ασχοληθήκαμε με διαφορετικούς τομείς, απασχοληθήκαμε σε διαφορετικούς τομείς στο Αφγανιστάν. Για το ιστορικό μου, ε, εκπαιδεύτηκα ως γλωσσομαθής αξιωματικός και εκεί με αυτά τα θέματα ασχολήθηκα στο στρατό. Οποιαδήποτε απορίες έχετε για τις γυναίκες στο στρατό, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Και εγώ είμαι ε, υπέρμαχος της ισότητας των γυναικών και στο στρατό, δηλαδή να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει από τις γυναίκες στο στρατό με τους άντρες, γιατί όπως κάποιος είπε, η ε, κυρία Γιανακουδάκη, αν δεν κάνω λάθος, που δυστυχώς έφυγε, η σφαίρα δεν κάνει διαφορά μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Και όταν κανείς έχει εκπαιδευτεί τόσο σκληρά όσο ένας άνδρας και γίνεται τόσο ισχυρός και δυνατός ως άνδρας, κερδίζει και το σεβασμό των ε, συναδέλφων. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι γυναίκε στο Αφγανιστάν είναι ε, ο πιο παραγωνισμένο ίσως πόρος αυτής της χώρας και θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να διαμορφώσουμε πρόσφορες συνθήκες για τη διευθέτηση αυτής της ε, σύραξης. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη σύραξη στον κόσμο. Όταν πρώτα να πάω στο Χέλμαντ, ε, έκανα διάφορε προκαταστήσει προκατακτικές καταρτήσεις και μάλιστα είχα συναντήσει και συναδέλφους άνδρες και όσο περισσότερο μιλούσα μαζί τους ε, ε, δημιούργησα την πεποίθηση ότι πρέπει να στείλουμε γυναίκες σε αυτό το πόλεμο γιατί εκεί είναι που είναι ιδιαίτερα καταπιεσμένες οι γυναίκες. Στο Αφγανιστάν βλέπετε ότι από το κράνος μου υπάρχει, βλέπουμε την αλογουρά μου και νομίζω ότι αυτή η εικόνα έμεινε εξίδηλα χαραγμένη στο μυαλό των γυναικών στο Αφγανιστάν. Η αλογουρά που βγαίνει από το κράνος. Μάλιστα ζήτησα να εργαστώ στο τμήμα ΣΥΜΙΚ, την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, με στόχο να επισκευάσουμε σχολεία, δρόμους όπου γίνεται να κατασκευάσουμε ε, γέφυρες και μάλιστα ήμουν η πρώτη γυναίκα σε τέτοια μονάδα πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και στην αρχή ο προϊστάμενός μου με ρώτησε αν θα μπορούσα να έρθω σε επαφή με μερικές γυναίκες στο Αφγανιστάν. Να τις βρω πρώτα, να βρω πού βρίσκονταν για να μιλήσω μαζί τους και όταν έφτασα επί τόπου το 2007, όταν πρώτα έφτασα στο Αφγανιστάν, ο Βρετανικός και ο Δανικός στρατός ήξεραν μόνο πέντε γυναίκες μέσα στο Χέλμαντ, ε, μία πόλη που αριθμεί ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Δύο εκατομμύρια στην ευρύτερη περιοχή και γνώριζαν μόνο πέντε γυναίκες. Και τις γνώριζαν γιατί δύο ε, Βρετανίδες ε, στρατιώτες ε, είχαν σε μια περιπολία πεζή γνωρίσει και πιάσει κουβέντα με δύο Αυγανές και κράτησαν και τα νούμερα των κινητών τους. Έτσι γνώρισαν τις πέντε γυναίκες και μάλιστα αυτή είναι η φωτογραφία της Κούλα Λέι, μιας καταπληκτικής γυναίκας που σήμερα νομίζω ότι έχει εκλεγεί και συμμετέχει σε επαρχιακό συμβούλιο στην πόλη του Γκερίσκ. Έχει εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος εκεί είναι μορφωμένη, μεσήλικη και χείρα και μάλιστα ε, η χειρία στο Αφγανιστάν είτε μπορεί να είναι ανυπόφορη αν δεν έχει κανείς πόρους ή και καταπληκτική γιατί είναι η και καταπληκτικη γιατι ειναι κυρια του αυτού της και μπορεί να, να λάβει τις αποφάσεις μόνη της. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα και ίδρυσε και ένα κέντρο για γυναίκες στο Αφγανιστάν που μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση. Βλέπετε πίσω αυτά τα γυαλιστερά, αυτές τις γυαλιστερές στολές που πάντα προσελκύει την προσοχή των γυναικών. Βλέπετε τις Αφγανές εκεί και μάλιστα σε συνεργασία με τη γυναίκα αυτή ξεκινήσαμε πολλά σχέδια με στόχο να βελτιώσουμε το προσωπικό εισόδημα, να δημιουργήσουμε κάποιες δεξιότητες και να μπορέσουν αυτές οι γυναίκες να βγάζουν λεφτά μόνες τους. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζουν και βγάζουν κάποια χρήματα, τότε αποκτούν και μεγαλύτερη ισχύ και εξουσία και εντός της οικογένειάς τους. Και ξεκινήσαμε διάφορα μικροσχέδια πτυνοτροφίας, μαθήματα ραπτικής, αλφαβητισμού, αγγλικών, ύφασης χαλιών. Δεν πέτυχαν βέβαια όλα αυτά τα σχέδια, αλλά πολλά από αυτά πέτυχαν, γιατί πραγματικά οι γυναίκες όταν αρχίζουν και βγάζουν χρήματα, τότε εγκαρδιώνονται, ενθαρρύνονται και έχουν και πολύ περισσότερα ενάυσματα για να συνεχίσουν. Αρχικά, όπως σας είπα, γνωρίζαμε γνωρίσαμε μόνο πέντε γυναίκες και μετά από τέσσερις μήνες παρουσίαση εκεί ε, γνωρίσαμε τουλάχιστον 500 γυναίκες. Ε, δηλαδή βλέπετε πόσο γρήγορη ήταν η εξέλιξη και όλο και περισσότερες γυναίκες ε, επιδίωκαν την επαφή. Αυτή εδώ είναι Φατιμά. Η Φατιμά φοράει μπουρκα, είναι πρωτότοκη σε μια οικογένεια μουλά, μουλάδων, σπούδασε, έγινε δασκάλα, ε, ξεκίνησε ένα σχολείο και μάλιστα συγκέντρωνε και χρήματα για να ιδρύσει σχολείο για κορίτσια και μάλιστα πρόσφατα συμμετείχε και στις εκλογές για το Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί της αντίπαλοι για να την, για να την εκφοβήσουν σκότωσαν τον σύζυγό της και δυστυχώς και ένας γιος της ε, σκοτώθηκε από στρατιωτικό όχημα σε ατύχημα. Δεν θα αναφέρω τι εθνικότητα ήταν το όχημα. Πάντω είναι μια πολύ ισχυρή γυναίκα, έχει φοβερή προσωπικότητα και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα δικαιωμάτων γυναίκας και ξέρει πραγματικά τι χρειάζονται οι γυναίκες και προσπαθεί να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις. Εδώ βλέπουμε τη Φάουσα Σίση που βρίσκεται εν μέσω πολλών παιδιών και είναι σημαντικό σημείο επαφή ε, για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν και πάλι του Αφγανικού Υπουργείου για τις γυναίκες. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί στο Αφγανιστάν αυτό που μετράει είναι ότι οι γυναίκες πέρασαν τόσο δύσκολα που χρειάστηκαν πραγματικά ένα σημείο επαφή ε, για, για τις επαφές τους με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και η, αυτή η ξεωματούχος επαφής είναι η Σάλμα. Και συνάντησα και εγώ πολλές γυναίκες που πραγματικά δεινοπάθησαν και πολλές φορές ε, η επαφή τους με στρατιωτικούς ε, δυσχεραίνει τη θέση του απέναντι στου Ταλιμπάν. Πολλοί Ταλιμπάν όταν βλέπουν ότι τέτοιε γυναίκε έχουν επαφέ με στρατιωτικού, με στρατιωτικό προσωπικό, κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή του. Είναι σημαντικέ πληροφορίε που λαμβάνουμε μένα από του άνδρε, αλλά όταν ξεκινούμε συζητήσει με γυναίκε, μαθαίνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα για τι κοινωνικέ δομέ, για τι φιλετικέ δομέ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μάθαμε ποια είναι τα όνειρά τους, οι προσδοκίες τους, ποια είναι η καθημερινότητά τους και η πραγματικότητά τους. Η UNIFEM ε, μας ενημέρωσε ότι 87% των γυναικών υφίστανται βία στο σπίτι τους. Και αυτό δεν έχει σχέση με τον πόλεμο, αυτό έχει σχέση με τις παραδόσεις στη, στο νότιο Αφγανιστάν. Και μάλιστα και εγώ έκανα κάποιες έρευνες και διαπίστωσα ότι στις ομάδες γυναικών ε, που συναντήσαμε, 70% των γυναικών αυτών ε, έζησαν βία στο σπίτι, είτε εις βάρος τους, είτε εις βάρος των παιδιών τους. Η συνομιλία με τις γυναίκες μας έδωσε μια νέα προοπτική και νέα σκοπιά για, το, για ποιο λόγο υπάρχουν ακόμη και συνεχίζουν το έργο τους, τη δράση τους οι Ταλιμπάν. Και μάλιστα βρήκαμε κάποιους τρόπους για να, τους κατα, να καταπολεμήσουμε την παρουσία τους στην κοινωνία. Βέβαια ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε φίλοι ελληνικοί ε, μετά την πρώτη μου περιοδία στο Αφγανιστάν ήρθα μεταφέροντας το μήνυμα των γυναικών του Αφγανιστάν που μου είπαν πείτε ευχαριστώ στις Δανέζες μητέρες που έστειλαν τα παιδιά τους στρατιώτες να πολεμήσουν στο Αφγανιστάν. Μπορεί σε μερικούς να μην ε, αρεστώ αυτό το μήνυμα, αλλά αυτή, αυτό ήταν το μήνυμα των γυναικών του Αφγανιστάν και αυτό και αποφάσισα και έγραψα και βιβλίο σχετικά, γιατί πολλά αρνητικά συνέβησαν στις γυναίκες εξαιτίας του πολέμου και συνέβη, αυτό και στο Αφγανιστάν, αλλά ε, δημιουργήθηκαν και ευκαιρίες στις ε, γυναίκες, ιδιαίτερα στο νότιο Αφγανιστάν που βρέθηκα εγώ και μερικές τις εκμεταλλεύτηκαν κιόλα. Μας είπαν στείλτε μας και γυναίκες στρατιωτίνες, γιατί για μας ε, είναι πολύ ενθαρρυντικό να σας βλέπουμε να περπατάτε με το πολυβόλο σας. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι και γυναίκες μπορεί να έχουν δουλειά και μάλιστα σκληρή δουλειά. Το είπα αυτό σε έναν άνδρα οδηγό και το έκανε για πλάκα. Ε, με χαιρετούσε κάθε φορά που έδινα διαταγή και μάλιστα προς μεγάλη τέρψη των γυναικών γιατί κάθε φορά που έβλεπα μια γυναίκα να διατάζει άντρες ε, πανηγύριζαν. Νομίζουμε ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στο Αφγανιστάν με τη θέση των γυναικών. Άρχισαν ε, οικειοθελώς να έρχονται και να βρίσκουν γυναίκες ε, δίνοντάς μου πληροφορίες για τους Ταλιμπάν. Βέβαια, οι γυναίκες είναι αυτές που θα βρεθούν χαμένες με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία γι' αυτό και ήρθαν και με βρήκα δίνοντας πληροφορίες για τους Ταλιμπάν. Αυτή η πανέμορφη γυναίκα είναι η ήταν μία από τις πληροφοριοδότησές μας, αλλά πολλές άλλες γυναίκες ε, συμμετείχαν στην παροχή πληροφοριών για τους Ταλιμπάν. Είχαμε στον Καρέσκ έναν βομβιστή αυτοκτονία που σκότωσε 42 ανθρώπου. Ήρθε μια γυναίκα και μου είπε πού είχε διαμείνει αυτό ο βομβιστή, ποιο τον βοήθησε, ποιο τον υπέθαλπε, ποιο του έδωσε όπλα, βόμβε, ποιο τον βοήθησε να φτάσει στον τόπο τη ε, βομβιστική αυτοκτονία. Και μάλιστα συγκέντρωσε όλες αυτές τις πληροφορίες ακούγοντας σχόλια από διάφορες γυναίκες στην πόλη. Γιατί οι γυναίκες μιλάνε, μιλάνε μεταξύ τους. Τέτοιες πληροφορίες λοιπόν κυκλοφορούν μεταξύ των γυναικών και ήταν σημαντική πηγή πληροφοριών για μας οι γυναίκες. Είχαμε μια άλλη περίπτωση όπου μια γυναίκα μας είπε πού φυλάγουν τα όπλα, ταυτότητε και τα λοιπά διάφορα στοιχεία και συγκεντρώσαμε τόσε πληροφορίες που στείλαμε ειδικά αποσπάσματα σε εκείνη την περιοχή και καταφέραμε να ε, εξαρθρώσουμε εκείνο το κύκλωμα. Λυπάμαι που σα τα λέω όλα αυτά, αλλά όταν μετέφερα τι πληροφορίε μου στο Δανικό και Βρετανικό στρατό και είπα ότι έχουμε έναν σύμμαχο στο Αφγανιστάν που τον είχαμε μελήσει μέχρι στιγμή, όλοι έπεσαν από τα σύννεφα, αλλά δεν είχαμε καμία επαφή μέχρι τώρα, τότε με τι γυναίκε, δεν καταφέραμε να ε, βγάλουμε κάποιε πληροφορίε από αυτέ. μετά καταφέραμε και αξιοποίησαμε αυτή την πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Μέχρι τότε τι αγνοούσαμε τελείω. Σε ό,τι αφορά την θέση των γυναικών στα θέματα ασφάλειας, είχα πολλές ε, και πολύ ωραίες συναντήσεις με γυναίκες. Κάποιος σύμβουλος μου ζήτησε να θέσω το ζήτημα του νομικού συστήματος ε, στο Αφγανιστάν και τι γνώμη έχουν οι γυναίκες γι' αυτό. Δεν χρειάζεται κανείς είναι για να φανταστεί ότι δεν ε, είναι και πολύ καλά τα πράγματα με το δικαιωτικό σύστημα του Αφγανιστάν. Πάντω, όταν είπε στι γυναίκε ότι θέλουν να μιλήσουμε για το σύστημα τη δικαιοσύνη, μου είπαν Α αφήσουμε αυτό το θέμα. Είναι διεφθαρμένο το σύστημα, δεν λειτουργεί, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν έχει καν νόημα να το συζητούμε γιατί ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Κατάφερα να τις πείσω να έρθουν μαζί μου παρά το, τη ματαιοπονία που πίστευαν ότι διέπραταν, γιατί τη έπεισε ότι μόνο να αρχίσουμε και μιλάμε για αυτό το θέμα μπορούμε να φέρουμε κάποια αποτελέσματα. Ε, ήρθαν λοιπόν στι συνεδρίε και πραγματικά θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η συνάντηση. Στην αρχή επικρατούσε ε, σιωπή. Κάποια στιγμή μια γυναίκα πήρε το λόγο και είπε ότι το πρόβλημα με εμά τι γυναίκε είναι ότι επειδή δεν έχουμε χρήματα δεν μπορούμε να δωροδοκίσουμε του δικαστέ για να έχουμε πραγματική δικαιοσύνη. Πραγματικά έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπο τον ήλιο με το σχόλιο αυτό και μα είπε και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα νερά κορίτσια που τι παντρεύουν σε ηλικία 8, 10, 12 ετών και δεν γνωρίζουν ότι είναι παράνομο κάτι τέτοιο. Γιατί ακόμη και ο Αφγανικό νόμο προβλέπει ω 18 την νόμιμη ηλικία γάμου. Αλλά δεν το γνώριζαν αυτό οι περισσότερε γυναίκε. Βέβαια, στην πράξη δεν θα άλλαζε και πολύ το θέμα, αλλά τουλάχιστον θα έδινε ένα επιχείρημα στι γυναίκε στη συζήτηση με του συζύγου του, προκειμένου να βάλουν τουλάχιστον αυτή την, αυτό το αναγκαστικό πάντρεμα, μέχρι να γίνει το κορίτσι τουλάχιστον 15, ώστε μετά την εγκυμοσύνη να έχει περισσότερε πιθανότητε επιβίωση. Δεν υπάρχουν γυναίκε δικαστίνε. Ε, δεν έχουν πρόσβαση καν στη δικαιοσύνη οι γυναίκε. Και το είπα αυτό και από την αρχή. Όταν επέστρεψα στο Αφγανιστάν ένα χρόνο μετά, διαπίστωσα ότι είχαν ξεκινήσει κάποιε ομάδε μελέτη ε, του αφγανικού δικαίου. Και αυτό έκαναν. Μελέτησαν όλε τι πτυχέ ε, του αφγανικού δικαίου που σχετίζονταν με δικαιώματα των γυναικών, δικαιώματα των παιδιών. Στη δεύτερη μου περιοδία στο Αφγανιστάν είχα παρόμοιες πρωτοβουλίες και παρόμοια σχέδια, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Συμμετείχα και σε άλλα πτυχές της, τη σύραξη του Αφγανιστάν. Τώρα έχουμε πέντε εκλεγμένες γυναίκες στο Επαρχιακό Συμβούλιο του Κεραίας και έχουμε τέσσερις γυναίκες σε άλλο Επαρχιακό Συμβούλιο. Και δεν είναι πια ε, ασυνήθιστο να συμμετέχουν γυναίκες στην πολιτική συζήτηση. Κάτι που ήταν σχεδόν αδύνατο όταν πρώτο πήγα στο Αφγανιστάν. Και έρχομαι στα συμπεράσματά μου ένα από του λόγου ε, που πιστεύω θα πρέπει να αναμίξουμε αυτέ τι γυναίκε είναι ότι ε, γιατί εντό τη οικογένειά του έχουν ε, εξουσία για λήψη αποφάσεων. Μπορεί στον δρόμο να μην τίποτα, μπορεί εκτό των τυχών τη οικογένεια να μην λένε τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που μια γυναίκα μπορεί να πείσει τον άντρα τη, έχει πραγματικά εξουσία στα χέρια τη. Έχουν πολλή επιρροή στι άντρε και κυρίω στα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Και πάνω από το μισό του πληθυσμού είναι κάτω των 25 ετών στο Αφγανιστάν. Ποιο θα μιλήσει με αυτά τα παιδιά, οι γυναίκε. Και οι γυναίκε μπορεί να μην έχουν άμεση πρόσβαση στη, στη λήψη αποφάσεων, αλλά έχουν άλλου τρόπους για να επηρεάσουν τα πράγματα και έχουν πραγματικά επιθυμία για κάτι τέτοιο. Μίλησα με πολλέ γυναίκε που μου είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα οι Ταλιμπάν θα με σκοτώσουν. Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με νοιάζει είναι το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δίνουν τη μάχη τους οι γυναίκες, για να έχουν καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους και έχουν οι ίδιες ε, εξουσία στην οικογένειά τους, έχουν βάρος στην οικογένειά τους. Και λυπάμαι που μακρηγορώ, αλλά ήθελα να δείξω στις γυναίκες ότι είμαστε στο πλευρό τους Τώρα, γιατί θέλουμε γυναίκες σε δυνάμεις ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα και η αστυνομία και ο στρατός είναι ο καθρέφτη του πληθυσμού. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα που έχει βιαστεί να μιλήσει με έναν άνδρα αστυνομικό. Αν μπει στο αστυνομικό τμήμα και βλέπει πέντε άνδρες, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα την πιστεύουν ότι κακοποιήθηκε ή ότι έπεσε θύμα βιασμού. Και γυναίκες λοιπόν θέλουμε στα, στις, στις, ομάδες, στις δυνάμεις ασφαλείας. Άλλωστε έχω την αίσθηση ότι οι γυναίκες ε, δεν είναι τόσο επιρρεπείς στη δωροδοκία, στη διαφθορά. Αυτό το λέω μόνο για το Αφγανιστάν. Και στη Μόσχα είχα περάσει ένα διάστημα και νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκε μία μονάδα 250 αστυνομικών γυναικών σε μοτοσυκλέτες γιατί διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες ήταν λιγότερο διεφθαρμένες και μάλιστα το 2005 όταν πέστρεψα, ο ο μεγαλύτερος φόβος του κόσμου τότε ήταν να μην τους σταματήσει η αστυνομία γιατί θα ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν ε, φακελάκι, να δωροδοκίσουν τον αστυνομικό πριν εμφανιστούν οι γυναίκες στην αστυνομία. Επίσης, όταν έχουν και γυναίκες σε μία μονάδα, οι άνδρες δεν πρόκειται να γκρινιάζουν, γιατί όταν βλέπουν τις γυναίκες ότι κάνουν μία δουλειά, δεν πρόκειται αυτοί ε, να μείνουν πίσω. Όταν με σταμάτησε ε, ένας Αφγανός ε, στρα, ε, ε, στρατηγός και με είδε 1,80 και, και οπλισμένη σαν αστακό, μου είπε θέλω γυναίκες σαν και εσάς. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όμως αρκετές, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε γυναίκες στο στρατό και έχουμε και πολλοί αξιόλογες αλεξιπτοτίστριες Ποια μαθήματα αντλήσαμε. Θα πρέπει να στείλουμε γυναίκες επί τόπου. Αν δεν στείλουμε γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν πρόκειται να εμπλέξουμε τον τοπικό πληθυσμό. Τις ντόπιε γυναίκε. Αδύνατον ένας Δανό στρατιώτη ε, να ξεκινήσει συζήτηση με μια Αφγανή. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αν είναι πολιτικό, εντάξει, έχει συνηθίσει να μιλάει με άνδρε. Αλλά μια, μια απλή γυναίκα δεν πρόκειται να μιλήσει με άνδρα. Θέλουμε λοιπόν συμβούλου ε, ε πληθυσμού, θέλουμε στρατιωτικού, θέλουμε αστυνομικού γυναίκε. Γιατί ωραία να μιλάμε για ισότητα, αλλά με το έργο μας θα πρέπει να δείξουμε ότι το εννοούμε. Και θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμε, στην προηγούμενη διαφάνεια για τις ένοπλες δυνάμεις. Πέρυσι, 18 Αφγανές ζήτησαν να μπουν στην αστυνομία στο Λέσκεβαρ, στην τοπική αστυνομία, ε, σε μια επαρχία του Χέλμαντ. 18 γυναίκες ε, Αφγανές βρήκαν το κουράγιο, είχαν τα κότσια να ε, υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στην αστυνομία. Αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένας κατερτισμένος σύμβουλος άνδρας για για να αναλάβει αυτό το έργο. Έχουν θάρρος, έχουν επιθυμία, έχουν ζήλο, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκαν μέντορες για να αναλάβουν την κατάρτισή τους στην αστυνομία. Λυπούμε, λυπούμε, γιατί υπάρχει επιθυμία, αλλά δεν υπάρχουν τα μέσα αυτή τη στιγμή. Σε μια χώρα σαν το Αφγανιστάν, σίγουρα τουλάχιστον μία γενιά θα χαθεί αν δεν κάνουμε κάτι. Υπάρχουν πολλές γυναίκες με πυγμή, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, γιατί πολλές φορές είναι εσωστρεφείς και φτύνουν να μυρολατρούν και να αποκαρδιώνονται. Θα πρέπει να τους ξαναδώσουμε κουράγιο, να τις επαναφέρουμε στο δρόμο και φυσικά να κάνουμε κάτι και για τους άνδρες, γιατί αν έχουμε μόνο σχέδια για τις Αφγανές γυναίκες θα ζηλέψουν τόσο πολύ οι άνδρες που θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν αυτά τα σχέδια και να μην καρποφορήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι και για τους άνδρες στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αν Κατρίν Ριευνίτσκι που μοιράστηκε μαζί μας ε, τις εμπειρίες σου στον τομέα αυτών. Θα ακούσουμε τώρα συναδέλφους που ασχολούνται με την εκθεσή πρωτοβουλίας. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην εκπρόσωπο του ΕΛΚ, την κυρία Νεντέλσεβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά πρώτα απ' όλα να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές αυτής της ακρόασης και τους προκεκλημένους που είχαν το θάρρος να προσεγγίσουν ένα θέμα που δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι και εξαιρετικά πολύπτυχο και περίπλοκο μας έδωσαν όμως πολλά στοιχεία για το ρόλο των γυναικών και της κοινωνίας γενικά σε θέματα σειράξεων. Ρίχνοντας μια ματιά στην αίθουσα, διαρωτόμαστε πού είναι το υπόλοιπο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Μακάρι να είχαμε περισσότερους άντρες στην αίθουσα να μου δώσουν και τη δική τους σκοπιά. Φυσικά δεν απευθύνομαι εδώ στους παρόντες, θα ήθελα να με ακούσουν οι απόντες επανέρχομαι στο θέμα των συνεπειών των σειράξεων στις γυναίκες. Είναι πολλές αυτές οι σειράξεις. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι γυναίκες έχαναν τους συζύγους τους στο μέτωπο και είδαμε διάφορα παραδείγματα από πολλές χώρες που έδειξαν ότι οι γυναίκες μπορούν να υποστούν αναγκαστικό εκτοπισμό, να φυλακιστούν, μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση που χωρίς κανένα πόρο πρέπει να αναλάβουν το νοικοκυριό μόνες τους. Άκουσα και ίσως την ε, χειρότερη συνέπεια των σειράξεων για τις γυναίκες που είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα και οι βιασμοί. Έχουμε φυσικά την ε, Σύμβαση 1325, το ψήφισμα του ΟΗΕ, που το ακούσαμε από την πρώτη προσκεκλημένη μας και την κυρία Μαν. Έχουμε πολλά ε, διεθνή κείμενα, συμβάσεις, ψηφίσματα που καταδικάζουν φυσικά τις βιοπραγίες και μάλιστα τα σεξουαλικά εγκλήματα των τελευταίων ετών πετύχαμε να χαρακτηριστούν ως εγκλήματα πολέμου. Αλλά βλέπουμε ότι οι βιασμοί είναι πολλές φορές ως ένα όπλο στον πόλεμο. Όταν λέμε πάντως εγκλήματα πολέμου εννοούμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται αυτά τα εγκλήματα και ως τρόποι εξευτελισμού, ταπείνωσης και εκφοβισμού. Βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματά τους και στα θύματα, αλλά και ε, πιο πέρα από αυτά. Για τα θύματα έχουμε τις σωματικές συνέπειες, αλλά έχουμε πρώτα απ' όλα τις ψυχολογικές συνέπειες, που είναι πολύ πιο επώδυνες και χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν. Όταν μιλούμε για τις ψυχολογικές συνέπειες, φυσικά υπάρχει το προσωπικό τραύμα, η κατάθλιψη. Αυτό όμως που ε, περισσότερο με σοκάρει είναι η απόρριψη του θύματος και η στιγματοποίηση του θύματος από την οικογένεια, από την κοινωνία. Οι γυναίκες ε, θεωρείται ότι έχουν ατιμαστεί και έτσι απορρίπτονται και από την οικογένειά τους και από το κοινωνικό τους περίγυρο. Γίνονται δύο φορές θύματα, λοιπόν, αυτό να μην το ξεχνούμε ο αντίκτυπος αυτός δεν αφορά τη γυναίκα μόνο ως θύμα. Ο αντίκτυπος αυτός είναι ευρύτερος και τριπλός θα έλεγα. Είναι αντίκτυπος προς τα παιδιά, είναι αντίκτυπος προς τους άνδρες, αλλά και αντίκτυπος για ολόκληρη την κοινωνία. Θα ασχοληθώ και με τις τρεις πτυχές. Ο αντίκτυπος στους άνδρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ίδιοι άνδρες θεωρούν ότι όταν μια γυναίκα υπέστη βιασμό, όταν υπέστη επίθεση, ε, δεν κατάφερε ο ίδιο να την προστατεύσει, δεν κατάφερε να προστατεύσει τη σύζυγό του, την οικογένειά του. Οπότε ταπείνωση αισθάνεται και ο ίδιο ο άντρα. και μερικέ φορέ αυτό ζητούν οι αυτούργοι, ακριβώ να αποκαρδιώσουν ή να εξευτελίσουν, να τιμάσουν και τον ανδρικό πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στα παιδιά, σε ορισμένε χώρε και θα σα δώσω το παράδειγμα τη δημοκρατία του Κογκό, θεωρούμε ότι οι, οι απόγονοι κυλιδώνονται από το βιασμό και πολλές φορές οι γυναίκες για να αποφύγουν κάτι τέτοιο προβαίνουν σε εκτρώσεις με αθυγιεινές συνθήκε είτε σκοτώνουν τα παιδιά τους κατά τη γέννηση. Τριπλός λοιπόν ο αντίκτυπος. Και υπάρχει και συνέπεια για ολόκληρη την κοινωνία. Θυμάστε τι έγινε τη δεκαετία του 90 στα Βαλκάνια ή στη, στον πόλεμο της, της Ρουάντα. Είχαμε είτε μαζικούς βιασμούς είτε αναγκαστικές ε, εγκυμοσύνες για λόγους εθνικής κάθαρσης η επόμενη γενιά λοιπόν είναι επίσης θύμα αυτής της κατάστασης. Σε περίπτωση ε, βιασμού ή αναγκαστικής εγκυμοσύνης ε, έχουμε το στίγμα που μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη και μια διαιώνιση των αποτελεσμάτων του πολέμου. Δεν περιορίζεται σε μια γενιά δηλαδή το τραύμα, αλλά συνεχίζεται και στις επερχόμενες γενιές. Πραγματικά είναι ζωφερός αυτός ο πίνακας των ε, συνεπειών των σεξουαλικών αυτών βιωτήτων και εγκλημάτων. Το θέμα είναι πώς ε, τα ισχύοντα μέσα που έχουμε και τους ισχύοντες μηχανισμούς θα τους καταστήσουμε πιο αποτελεσματικούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είναι πολύ εύστοχα αυτά που μας είπατε. Στα πλαίσια των λύσεων μπορούμε να αναζητήσουμε τις λύσεις σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο κρατικό και στις στρατιωτικές δομές, σε επίπεδο κοινωνικό, εδώ πολύ σωστά επισημάνθηκε ο ρόλος του σχολείου και της διαπαιδαγώγησης και σε προσωπικό επίπεδο, στο επίπεδο των γυναικών. Όταν μιλούμε για το κρατικό επίπεδο, πρωταρχική ευθύνη του κράτους είναι να εξασφαλίσει την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας από τις ε, ε, δικαστικές αρχές. Όλες οι χώρες σχεδόν έχουν τη σωστή νομοθεσία, έχουν όλες επικυρώσει τα διεθνή, τα διεθνή κείμενα, τις διεθνείς συμβάσεις, απλώς θα πρέπει να τις εφαρμόσουν, να αισθάνονται εμπιστοσύνη οι γυναίκες στην δικαιική τάξη. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο στρατό, σίγουρα θα πρέπει να προβλέψουμε ανάλογες ποινές για τέτοιες δράσεις. Οποιοδήποτε αυτούργος, είτε είναι στρατητικός είτε παραστρατητικός δεν θα πρέπει να υπολογίσει την ατιμορρησία τέτοιων πράξεων. Γιατί μερικές φορές ε, οι επίδοξοι βιαστές γνωρίζοντας ότι ή προσβλέποντα την ατιμορρησία δεν διστάζουν να πραγματοποιήσουν το έγκλημα. Ενώ αν είχαμε ανάλογες αυστηρέ ποινέ, θα λειτουργούσαν εκφοβιστικά. φορέ φορές στρατιωτικέ δυνάμεις ε, λένε οι χώρες ε, εκφεύγουν του ελέγχου τους. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού, γιατί οι γυναίκε εκεί ανήκουν. Θα πρέπει να ελεγχθεί το στρατιωτικό προσωπικό. Επίση, οι κοινότητε που περιβάλλουν τι γυναίκε θα πρέπει να προσπαθήσουν να αφυπνίσουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τις βιοπραγίες αυτές που γίνονται στις γυναίκες, ώστε το στίγμα και η απόρριψη να περιοριστούν. Πήγα πέρυσι στη Δημοκρατία του Κονγκό και είδαμε, είδα στις διάφορες πλατείες ε, είτε ε, ζωγραφιές που εξηγούν με απλό τρόπο τη, τα δεινά που υφίστανται οι γυναίκες από τέτοιου είδους σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Νομίζω ότι αυτό έχει διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα και στο Κιβού με διάφορα χορευτικά, με θέατρο για να μην προσβληθεί η ευαισθησία της παραδοσιακής κοινωνίας, προσπαθούν με τέτοιο πιο ήπιο τρόπο να διαπαιδαγωγήσουν τον κόσμο και να βελτιώσουν τη θέση της γυναίκας, ιδιαίτερα που έχει υποστεί τέτοιες επιθέσεις, τέτοια σεξουαλικά εγκλήματα. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει οι γυναίκες να αισθανθούν εμπιστοσύνη και να ενεργοποιηθούν, να γίνουν δραστήρια, δραστήριοι φορείς αυτής της αλλαγής και εμείς δεν μπορούμε παρά να τις εθαρρύνουμε. Ευχαριστώ κύριε Ναντέλσεβα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φιγερέιδο από ε, την ε, ομάδα Ενωμένη Αριστερά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Eh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες τις παρεμβάσεις τις διάφορες αναλύσεις που ακούσαμε και τις πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικές εμπειρίες ε, επιτόπου για τις προσπάθειες που έγιναν για τη βελτίωση των βιωτικών συνθήκων των γυναικών και την ανάμειξη των γυναικών στην ε, καταπολέμηση της ε, οικονομικής τους εξάρτησης και στη βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου γιατί πραγματικά αυτή η κατάσταση είναι, δίνει μια γυναίκα που εξαρτάται οικονομικά, είναι υποτελής και υφίσταται πολύ πιο εύκολα διάφορες επιθέσεις, όχι μόνο σε καιρό πολέμου, αλλά δυστυχώς και σε καιρό ειρήνης. Είναι σημαντικό λοιπόν οι γυναίκες να ανακτήσουν αυτή την ανεξαρτησία. Χαίρομαι για την πρόταση αυτή να εμπλακούν όλο και πιο ενεργά οι γυναίκες και εγώ πιστεύω ότι η δική μας συμβολή ε, ως γυναικών θα πρέπει να είναι σε επίπεδο πρόληψης του πολέμου, υπέρ της ειρήνης δηλαδή. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος δημιουργεί μια σειρά συνεπειών, όπου τα αρχικά του θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και άλλα θύματα, οι νεκροί για παράδειγμα που είναι και άνδρες και γυναίκες αλλά τις πιο σοβαρές συνέπειες ε, των σειράξεων τις φέρουν οι γυναίκες και τα παιδιά και εξαιτία ε, των ε, σεξουαλικών εγκλημάτων, των βιασμών αλλά πολλές φορές έχουμε παιδιά που γεννιούνται από τέτοια εγκλήματα και που γίνονται θύματα αυτής της κατάστασης με πολλούς και διάφορους τρόπους. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ειρήνη εμείς ως γυναίκες και να δούμε πώς μπορούμε να επέμβουμε για να αποτρέψουμε τον πόλεμο, να αποφύγουμε τη σύραξη. Και όχι απλώς να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες ή να κατευνάσουμε τις ε, συνέπειες ε, των θυμάτων του πολέμου. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο πρόληψης και αποτροπής θα πρέπει να δώσουμε το βάρος. Οι γυναίκες είναι το, αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό και ο ρόλος του στην κοινωνία θα πρέπει να είναι πιο εμφανής. Και μάλιστα οι γυναίκες κατά πάσα πιθανότητα είναι και πιο ευαίσθητες απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Οπότε, αν καταφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση να παρεύουμε σε επίπεδο διαπαιδαγώγηση λοιπόν υπέρ της ειρήνης σε διάφορους τομείς όπου έχουμε τέτοια δυνατότητα επέμβασης, νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει είτε σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο κυβερνητικό, είτε σε επίπεδο θεσμικό, κοινοτικών οργάνων, να, να επιμείνουμε στην ανάγκη διαπαιδαγώγησης της ειρήνης. Και νομίζω ότι τα σχολικά θρανία είναι ο χώρος που θα πρέπει να γίνεται πρώτα απ' όλα αυτή η διαπαιδαγώγηση. Θα πρέπει να έχουμε εκεί στα σχολεία σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ειρήνη. Έχουμε διεθνεί συμβάσεις, διεθνέ δίκαιο, έχουμε τις συμβάσει του ΟΗΕ και πολλές άλλες συμβάσεις και νομικά μέσα που μιλούν για συνεργασία αναπτυξιακή, για την ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών και ισότητα δικαιωμάτων όχι μόνο μεταξύ των δύο φύλων, αλλά ισότητα δικαιωμάτων σε πολλούς τομείς. Ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ των λαών και μεταξύ των χωρών, ώστε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Να έχουμε μια ανάπτυξη που θα δίνει περισσότερη προσοχή στον άνθρωπο, ώστε πραγματικά να μειωθεί η πείνα, η εξαθλίωση, να διαφυλαχθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, η πρόνοια, η υγεία, η παιδεία για όλους. Γιατί εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία και την ανάπτυξη. Και φυσικά σε επίπεδο κρατών και κοινοτικών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στη διπλωματία. Γιατί μέχρι στιγμής οι άνδρες ήταν κυρίως υπεύθυνοι για τις δημοκρατίες και τους πολέμους. Δεν λέω ότι οι γυναίκες είναι τελείως άμυρες ευθυνών, αλλά πρώτα απ' όλα οι άνδρες μέχρι στιγμής είχαν τα ενία της εξουσίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε καλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε ηθήνουσες θέσεις, σε ηγετικέ θέσεις και να ενισχύσουμε το ρόλο της διπλωματίας πριν καταφύγουμε στην πιο άμεση και ριζική απάντηση που είναι η κήρυξη του πολέμου. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δι... κανονίσουμε διαφορές. Δεν χρειάζεται να προσφεύγουμε στον πόλεμο και να δώσουμε σε αυτό έμφαση, στην πρόληψη, στην αποτροπή του πολέμου, στην αναζήτηση άλλων τρόπων διευθέτησης των διαφορών. Νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση όλες οι γυναίκες που ασχολούμαστε με την πολιτική. Χαίρομαι για αυτά που ακούσαμε για το Αφγανιστάν και την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών. Γιατί όμως αυτά δεν μας τα λέγατε πριν τον πόλεμο, γιατί δεν τα κάναμε όλα αυτά, όλη αυτή τη ε, συμμετοχή σας εκεί στην τοπική κοινωνία δεν τα, δεν κάναμε πριν από τον πόλεμο, ώστε να είχαμε αποφύγει όλη αυτή την καταστροφή, όλο αυτό τον όλεθρο, την εξαθλίωση, τους θανάτους, ακόμη και των γυναικών και των παιδιών. Υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για να αποφύγουμε τον πόλεμο, επαναλαμβάνω και επιμένω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φικερέιδο. Θα ακούσουμε τώρα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από την Κατερίνα Λέιρονεν που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σου δίνω το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί συνεχώ τα θέματα αυτά πολύ υψηλά στις προτεραιότητές του ε, και το εκτιμούμε ιδιαίτερως. Προσφάτως ε, άκουσα την κυρία Μάργκοτ ε, Βάλστρο, η οποία επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια παρέμβαση. Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί της και μίλησε και με τους 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ωραία συνεδρίαση και την εκτίμησαν ιδιαίτερα όλη την παρουσίαση της εκεί και ενδιαφέρονταν όλοι για τη συζήτηση με την κυρία Βάλστρομ. Νομίζω ότι έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συχνά δηλαδή διοργανώνουμε συνεδριάσεις επί του θέματος ε, και απλώς ε, έρχονται γυναίκες ε, και άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα δεσμευμένοι σε αυτά τα θέματα. Ε, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε την στρατηγική μάρκετινγκ και την αλλαγή της ορολογίας μας. Να αρχίσουμε να μιλάμε ε, για τις γυναίκες στην ασφάλεια ή για γυναίκες και άνδρες ε, και την ειρήνη και την ασφάλεια. Κάποια γρήγορα σχόλια για τις ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε. πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, όπως ενδιαφέροντα ήταν και τα σχόλια από την κυρία, συγγνώμη που θα προσφέρω λάθος το όνομά σας, ελπίζω να το πω σωστά, την κυρία Ριμπνίτσκι. Τα ίδια ακούμε και από τους εμπειρογνώμονές μας που είναι υπεύθυνοι στις αποστολές και στις επιχειρήσεις για τα θέματα φύλου. Κάποια από τα θέματα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η συμμετοχή των γυναικών. Μήπως τις θέτουμε σε κίνδυνο. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό όταν λαμβάνουμε εμπιστευτικέ πληροφορίες ε, και είναι γνωστό ε, κατόπιν ότι διαβιβάζουν τις πληροφορίες, ε, ε, μήπως τις θέτουμε σε κίνδυνο. Ε, παρά τα όσα ακούσαμε από τους συμβούλους μας σε θέματα αυτά, ε, ιδίω στο Τσάντ, ε, καταλαβαίνουμε σύμφωνα με αυτούς να έχουμε μια πλήρη εικόνα όταν λαμβάνουμε στοιχεία και από τους άνδρες και από τις γυναίκες από τις συμβούλους και για το ΝΑΤΟ και για τη δική μας ε, ε, αποστολή στο Αφγανιστάν. Μάθαμε ότι και οι άνδρες μπορούν να μιλήσουν με γυναίκες στο Αφγανιστάν και είχαμε και κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα από αυτή τη ε, συζήτηση επίσης. Εγώ δεν είμαι πυρογνώμων σε θέματα του Αφγανιστάν, απλώς λέω ότι μπορεί να ερίζουν και λίγο οι απόψεις επί του θέματος. Το να κάνουμε κάτι και για τους άνδρες επίσης. Ναι, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι συμμαχοί μας και να συμμετέχουν επικοδομητικά στην όλη διαδικασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το Κονγκό, όπου υπάρχει μια αστυνομική αποστολή στην Κόμα, στο Βόρειο Κίβο, με μια ομάδα που ασχολείται με τη σεξουαλική βία και εκπαιδεύει την τοπική αστυνομία η οποία αστυνομία στη συνέχεια εκπαιδεύει την αστυνομία του Κονγκό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο στρατηγικό στοιχείο, οι άνδρες επιτόπου να ε, εκπαιδεύουν τους άνδρες επιτόπου με τη δική μας υποστήριξη. Σήμερα Έχουμε προχωρήσει πέραν ε, της ε, απλής συνεργασίας και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το πρόγραμμα δράσης του 2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φύλλο και την ε, συμμετοχή των γυναικών ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έγγραφο για να το σχολιάσω ολόκληρο. Απλώς να σταθώ σε ένα σημείο και να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα έγγραφο που καλύπτει και την ευρωπαϊκή κοινότητα και την βοήθεια από πλευράς ευρωπαϊκής κοινότητας αλλά και την βοήθεια από πλευράς κρατών μελών. Επί παραδείγματι στις χώρες εταίρους γίνεται καταμερισμός εργασίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα μπορεί να είναι επικεφαλής ε, και ένα κράτο μέλο ε, σε θέματα φύλου στι χώρε εταίρου. Επιπλέον, διαθέτουμε και 70 περίπου σημεία επαφής στην αντιπροσωπεία μας που ασχολούνται συγκεκριμένα με το θέμα του φύλου. Ε, δεν στοχεύουμε σε θέματα προβολής. Ε, να σας πω όμως ένα ανέκδοτο. Αυτή τη στιγμή στην Τινησία υποστηρίζουμε τις γυναίκες για να είμαστε βέβαιοι ότι οι πτυχές του φύλου και τα θέματα των γυναικών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στις μεταρρυθμίσεις. Οι γυναίκες αυτές δεν θέλουν απαραίτητους προφανή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχουν ισλαμιστικές ομάδες που τις κατηγορούν ότι τις εκμεταλλεύεται ο δυτικός κόσμος. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να επιδείξουμε και τη δέωσα τακτική και μπορεί να μην προβάλλεται το έργο μας όσο θα θέλαμε να προβάλλεται. Θα θέλαμε να προβάλλουμε την υποστήριξη που παρέχουμε στις γυναίκες στην Τινησία, αλλά ε, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι δεν θα πρέπει πάντα να φαινόμαστε ότι υποστηρίζουμε τα θέματά τους να σας ε, επισημάνω και μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία και χαιρετίζω από την, ε, ε, το Τμήμα Πολιτικής, Εξωτερικής Πολιτικής, ένα έγγραφο για την εφαρμογή του 2035. Ασχολούμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιε είναι οι δεσμεύσει για την ευρωπαϊκή πολιτική και ότι το, από το 2008 υπάρχει μια συνολική προσέγγιση στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις, ε, τα ψηφίσματα 1325 και 1820. Έχουμε πλήρη τεκμηρίωση για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα στοιχεία αυτά στις αποστολές και στις επιχειρήσεις μας και να σας υπενθυμίσω και τις κατευθυντηρίες γραμμές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη βία κατά των γυναικών. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε και τον ε, τους όρους για ενδιαφέρουσες ε, περιφερειακές ε, ε, εκστρατείες για τη συμμετοχή των γυναικών κυρίως στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτά θα παρουσιαστούν αργότερα στο τέλος του έτους και στις αρχές του επομένου θα ήθελα να επικεντρωθώ για λίγα λεπτά σε κάποιες πιο πρόσφατες πληροφορίες. Μπορεί να γνωρίζετε ότι πέρσι, για παράδειγμα, υιοθετήσαμε δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνη και την ασφάλεια και τις γυναίκες. Όταν ε, ετοιμάσαμε την πολιτική του 2008 γνωρίζαμε ότι πρόκειται για ένα μικρό πολιτικό άνοιγμα. Δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνει τόσο εξαιρετική δουλειά όπως η Φιλανδία που αναφέρει και εδώ ότι είχε το καλύτερο πρόγραμμα δράσης. Δεν είχαμε χρόνο να σταθούμε στους δείκτες, τους ε, εκπονήσαμε αργότερα και αυτοί υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο πέρσι. Το Μάιο φέτος είχαμε και την πρώτη βασική έκθεση για τους 17 αυτούς δείκτες. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω κάποια από τα βασικά αποτελέσματα και κατόπιν θα ολοκληρώσω με κάποιες διαπιστώσεις και κάποιες συστάσεις επί τη βάση κυρίως αυτής της έκθεσης που είναι ένα δημοσιοποιημένο έγγραφο το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Καταρχάς, να σας πω ότι είχαμε πολύ καλό ποσοστό απαντήσεων, 24 από τα 27 κράτη-μέλη απάντησαν, όλες οι αποστολές ε, και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων απάντησαν. Είχαμε και 60% αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απάντησαν και ε, σταθήκαμε μόνο σε όσους βρίσκονται σε ε, περιοχές και σε επικίνδυνες χώρες. Ε, και λάβαμε και απαντήσεις από τους ειδικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας για τις γυναίκες σε πολλές χώρες, 75 τον αριθμό, Επομένως, ε, αναλαμβάνονται δράσεις ε, περίπου παγκοσμίως για ένα πολύ μεγάλο φάσμα δράσεων που ε, περνούν από την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων δράσης, όπου υπάρχουν εθνικά προγράμματα δράσης, ε, χρηματοδότηση σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνία των παλετών και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, συνδρομή και έγγραφο πολιτικής σε κυβερνητικές ε, δομές και ούτω καθεξής. Το βασικό μέσα που χρησιμοποιούνται από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης... είναι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι μη κυβερνητικοί φορεί και οι Τοπικές Αρχές ε, για την ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν αναφέρθηκε πολύ ε, το θέμα της ε, βοήθειας για τα μέσα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει και μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση επί του θέματος, αλλά μόνο τρεις αντιπροσωπείες αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Ε, υπάρχουν πολλά όμως ενεξελίξει στο πρόγραμμα δράσης ε, για φέτος, ε, για τα μέσα, για τη σταθερότητα. Επίσης προσμετρήσαμε και την πολιτική δράση, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική ως εργαλείο. Οι γυναίκες, η ασφάλεια και η ειρήνη έχουν συστηματικά συμπεριληφθεί στον ε, διάλογο με την Αφρική και στα ε, στους επόμενους μήνες θα οργανώσουμε και ένα σεμινάριο χαρτογράφησης για την ε, ε, προγράμματα που έχουμε στην Αφρικανική και Ευρωπαϊκή Ήπειρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε την δουλειά που κάνουμε στην Αφρική και θέλουμε να προχωρήσουμε και τις δράσεις για του, όσους διατηρούν την ειρήνη στην περιοχή της Αφρικής. Και φυσικά προχωρούμε και μέσω της ευρωμεσογειακής ετορικής σχέσης ε, στα προγράμματα δράσης της Κωνσταντινούπολης και του Μαρακές και συστηματικά Έχουμε συμπεριλάβει και συζητήσεις ε, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια με χώρες όπως είναι ο Καναδάς φυσικά που είναι ε, περίπου ταυτόσιμες οι απόψεις του με εμά, αλλά όπως επίσης και με χώρες όπως το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Παππούα Νέα, την Νότια Αφρική, τη Σομαλία, το Σουδάν και την Ουγκάντα. Θα πρέπει λοιπόν να διορθεί αυτή η πολιτική όθηση σε όλο το φάσμα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι έχουν δαπανίσει ε, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και το 2010 για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γυναίκες στην ασφάλεια και την άμυνα και αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα γιατί δεν απάντησαν όλα τα κράτη-μέλη και δεν έχουμε λάβει όλες τις πληροφορίες για την ανθρωπιστική βοήθεια ε, και σίγουρα το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε περίπου το 25% της υποστήριξης πήγε στο Αφγανιστάν βάσει της έκθεσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένο και θα ήθελα να κάνω μια σύσταση εδώ. Θα πρέπει να υπάρξει και μια ανάλυση αντικτύπου και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στο Αφγανιστάν γιατί είναι τόσο μεγάλη χρηματοδότηση αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης κρίσης και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μέσω ΝΑΤΟ. Ένα άλλη μεγάλη συνεισφορά είχαμε στην ε, περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής, ε, το Νεπάλ και τις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές. Επίσης έχουμε κάποιους δείκτες για τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές ε, γυναικών και φίλου. Εδώ τα στοιχεία είναι λιγότερο ενθαρρυντικά, διότι τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ανέφεραν ότι η υποστήριξη σε διαπραγματεύσεις είναι με άτυπο ή επίσημο τρόπο σε πολλές χώρες, αλλά πολλοί από αυτόν δεν μπορούσαν να μας πούν αν υπήρχε παρουσία γυναικών. Υπό την έννοια ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν αποτελούσε μία από τις επιτυχίες που τους ενδιαφέραν ιδιαίτερα. Και δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη έκθεση που έγινε, ελπίζουμε ότι αν ε, εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό μέσω των δικτών, θα μπορέσουμε ίσως να το προωθήσουμε περαιτέρω. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό σημείωμα για τη διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις με πολύ ενδιαφέρουσες δεσμεύσεις για το ρόλο των γυναικών, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως, ιδίω ε, δεδομένου ότι υπάρχει και ειδικό τμήμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα θέματα αυτά. Η εξαίρεση που αναφέρθηκε ήταν η Ουγκάντα, όπου οι γυναίκες σε επίπεδο κοινότητας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Τώρα, οι γυναίκε ω επικεφαλής αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αποστήλαμε τα ερωτηματολόγια στι 36 χώρε που καλύπταμε, υπήρχε μόνο μία γυναίκα επικεφαλής αντιπροσωπεία. Θα γνωρίζετε βεβαίω ότι είπα ότι εκπρόσωπος η κυρία Άνστον έχει επιτελέσει κάποια πρόοδο επί του θέματος και από τους τελευταίους διορισμούς που είχαμε έχουμε 9 γυναίκες επικεφαλής των αντιπροσωπιών και έχουμε φτάσει πλέον στις 26 γυναίκες. Ε, είναι διπλάσιο το ποσό από τα προηγούμενα στοιχεία και εξ όσο γνωρίζω η τάση είναι συνεχής και θα υπάρχουν και άλλοι σχετικοί διορισμοί ε, από την το εκπρόσωπο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό γυναικών ε, επικεφαλής ε, διπλωματικών ε, αποστολών ήταν 18% από τις απαντήσεις τουλάχιστον που λάβαμε. Το υψηλότερο ποσοστό είναι στη Σουηδία με 34%, Φιλανδία 33% και Εστονία 25%. Όμως ο μέσος όρος γυναικών σε αποστολές ασφάλειας και άμυνας ήταν 10%. 26 για τη Σουηδία, 16 για την Εστονία, ε, και μια ε, χώρα ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα στις αποστολές αυτές. Στις ειρηνευτικές αποστολές η συμμετοχή των γυναικών ήταν μόνο 5%. Επομένως τα στοιχεία ήταν λίγο καλύτερα από τι ε, ειρηνευτικέ αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, κάποια συμπεράσματα. Έχουμε λίγα πράγματα για ε, οφείλω στις ε, κοινέ δράσεις του Συμβουλίου που καθορίζουν τις αποστολές και τις επιχειρήσεις μας. Μόνο σε δύο κοινέ δράσεις υπήρχε συγκεκριμένη διατύπωση. Δεν αναφέρομαι στη σεξουαλική βία γιατί δεν τη θεωρώ ως ε, υποκατάστατο της γλώσσας που αναφέρεται στο φύλλο. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχώρησαν οι αποστολές στο έργο αυτό και σε όλες τις αποστολές υπήρχε και ε, σημαντική ε, αναφορά στα θέματα αυτά στα επιχειρησιακά έγγραφα. Επίσης, ε, οι χώρες μέλη ρωτήθηκαν αν υπάρχουν εθνικά προγράμματα δράσης για το 2025 και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερο. Τώρα, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, μόνο τέσσερις μας είπαν ότι καλύπτουν σχετικές πτυχές στις εκθέσεις τους ε, για τις γυναίκες. Ε, θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Μια πολύ σημαντική ε, έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή των ε, Μεγάλων Λιμνών που ήταν και υπέρμαχος της εφαρμογής του 2025. Ε, ελάχιστες γυναίκες ε, συγγνώμη, ελάχιστοι άνδρες εκπαιδεύονται για θέματα γυναικών, είναι γυναικείο το θέμα και εκπαιδεύουμε κυρίως γυναίκες και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Υπάρχουν και πολύ σημαντικές πρακτικές οι οποίες προέκυψαν και εξελίσσονται και ελπίζω μέσω της δημοσιοποίησης που έχουμε πλέον ε, να μπορέσουμε και να τις γνωστοποιήσουμε και να μπορέσουμε να τις γνωστοποιήσουμε ακόμα περαιτέρω. Στο Νεπάλ υπήρχε μια ομάδα τοπικού συντονισμού για το 2025 το οποίο είχε ως αποτέλεσμα και τη έγκρισης ε, του Εθνικού Προγράμματος Δράσης του Νεπάλ. Στη Σομαλία έγινε μια αξιολόγηση για τις δυνατότητες όλων των Υπουργείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά ψηφίσματα και εντοπίστηκαν προκλήσεις, δυνατότητας και σημεία εισόδου. Επιπλέον στη Σομαλία υποστηρίξαμε στη συγκέντρηση των φωνών των γυναικών για την έκθεση ε, γονιμότητας η οποία θα δημοσιοποιηθεί αργότερα και τα, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί ακούσαμε τι είχαν να πούν οι γυναίκες για το πώς αντιμετωπίστηκαν τα θέματα των γυναικών στη Σομαλία. Υπήρχε και σημαντικός εξορθολογισμός ε, για τα θέματα του φύλου στο Πακιστάν. Ε, περιλαμβάνεται τώρα σε πέντε πυλώνες της διαδικασίας και υπήρχε και μία πρωτοβουλία διασταυρούμενης ε, διαπαιδαγώγησης ε, στο Ανατολικό Τιμόρ, στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόνε και ε, ζητήθηκε να ετοιμαστούν και προγράμματα δράσης για το 1325. Υπήρχαν χώρες που υποστήριζαν συγκεκριμένες χώρες όπως για παράδειγμα η Φιλανδία, την Κένια. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, όπως για παράδειγμα την ε, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και ε, προσλήψεων. Και επίσης υπήρχε και μια συγκεκριμένη δήλωση ε, για το φύλλο που αναφέρονται στην αποστολή της UPOL COPS στην Παλαιστίνη, όπου υπήρχε και υποστήριξη από την τοπική κυβέρνηση. Ένα-δυο πράγματα να πω ακόμα. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μια στεναρή πολιτική και δεν είναι το πρόβλημα η πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κενά στην εφαρμογή, κυρίως επιτόπου. Το πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να εφαρμοστεί η πολιτική συστηματικά επιτόπου μέσω των επικεφαλής ε, των αντιπροσωπιών σε όλες τις αποστολές. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και νομίζω ότι είναι υπέρμαχος αυτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα πλήρες τμήμα ε, που ασχολείται με θέματα ε, φύλου στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Υπάρχει απλώς προσωπικό που από καιρούς καιρών ασχολείται με τα θέματα αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερα ε, σε θέματα χρηματοδότησης ε, και ε, ζητήσαμε από την Επιτροπή Προγράμματος Δράσης να έχει θέματα φύλου πριν καθορίσει τα έγγραφα πολιτικής για κάθε χώρα και νομίζω ότι αυτό είναι αισιόδοξο και θα πρέπει οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών να είναι υπόλογοι και να λαμβάνονται υπόψη συστηματικά τα στοιχεία αυτά. Στο πρόγραμμα δράσης για το φύλλο έχουμε δεσμευθεί και στην κατάρτιση όλων των επικεφαλείς των αντιπροσωπιών για τα θέματα φύλου. Το 2012 θα συνεχίσουμε τις εργασίες και να εφαρμόζουμε κάποιες νέε πρωτοβουλίε και την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε και με την αναθεώρηση της πολιτικής για να δούμε πώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν οι πολιτικές μας τις πιο πρόσφατε, εξελίξεις, πιο συγκεκριμένα τα όσα αφορούν τις ε, 1960 και 1889 τα ψηφίσματα αυτά για την ε, ε, ειρηνευτική διαδικασία και έχουμε και μια διαδικασία χαρτογράφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης ε, μοντέλα κατάρτισης τα οποία αφορούν το προσωπικό μας για θέματα φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας των παιδιών και έχουμε οργανώσει και συντονισμό μεταξύ των συμβούλων σε θέματα φύλου. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μία πρωτοβουλία Ισπανίας-Ολλανδίας για μαθήματα μίας εβδομάδας ε, σε κατάρτιση που βασίζεται σε διάφορες εναλλακτικέ εκδοχές και το πρώτο, ε, ε, ο πρώτος κύκλος μαθημάτων γίνεται αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη. Έχουμε εξετάσει και θέματα φίλου στη Λευκορωσία που έχει αναλάβει ε, την εκπόνηση βασικών δικτών και ένα, μία από τις υποκατηγορίες των δικτών του Πεκίνου είναι τα θέματα φύλου και ελπίζω να έχουμε υποστήριξη από το Ινστιτούτο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στους συναδέρφους ε, εάν έχουν να θέσουν ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Η κυρία ε, Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των ε, γυναικών στο Αφγανιστάν, που είναι μια χώρα που γνωρίζω αρκετά καλά. Η χώρα αυτή βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση δεκαετίες ολόκληρες από την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης με διαφορετικούς τρόπους ε, και διαφορετικές μορφές είχαν οι πόλεμοι αλλά δεν σταμάτησαν. Από το 2001 είμαστε κι εμείς εμπλεκόμενοι σε αυτή την παρέμβαση και μάλιστα το 2001 προβάλαμε αυτό το πόλεμο στην ε, ευρωπαϊκή κοινή γνώμη επιμένοντας σε αυτή την ανάγκη να πολεμήσουμε για να σώσουμε τις γυναίκες του Αφγανιστάν. Έτσι το προβάλαμε στην ε, κοινή γνώμη και αυτά τα επιχειρήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Εγώ γνωρίζω τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, έχω πολλούς δεσμούς με ενώσεις γυναικών στο Αφγανιστάν όλος παραδόξως ε, ανησυχούν τα μάλα αυτή τη στιγμή γυναίκες στο Αφγανιστάν ε, γιατί ξέρουν ότι διεξάγονται ελληνευτικέ διαπραγματεύσεις και η προοπτική αυτή τη ειρήνη που ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται με, ότι με διακριτικό τρόπο προετοιμάζεται πρόσφατα στην Γερμανία οι δύο τη εκπρόσωποι της, των ΗΠΑ συνάντησαν τον το εκπρόσωπο του Μουλά Ομάν. Αυτό δεν προβλήθηκε πολύ και στην συνδιάσκεψη του Λονδίνου οι ενώσεις ε, γυναικών του Αφγανιστάν διαμαρτυρήθηκαν και ε, έκαναν απεύθυνα διάβημα προς την ε, Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Κλίντο λέγοντας και με εμάς τι θα γίνει. Φοβούνται οι γυναίκες του Αφγανιστάν ότι θα είναι τα θύματα αυτής της διαπραγμάτευσης για την αποχώρηση των δυτικών, γιατί Ξέρουμε ότι οι δυτικέ δυνάμει το μόνο που επιθυμούν διακαβώ είναι να φύγουν από το Αφγανιστάν το συντομότερο δυνατόν. Αυτό φοβούνται λοιπόν οι γυναίκε του Αφγανιστάν, ότι θα μείνουν οι παραμελημένε αυτή τη κατάσταση και όταν θυμόμαστε τι επενδύσει που κάναμε στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα για τι γυναίκε, νομίζω ότι φέρουμε τεράστια ευθύνη στη χώρα αυτή, ιδιαίτερα απέναντι στι γυναίκε αυτή τη χώρα. Δεν έχω ούτε λύση, ούτε συγκεκριμένη απάντηση, ούτε είμαι φιλοπόλεμη, ούτε είμαι υπέρ τη συνέχιση του πολέμου. Δεν εννοώ αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουμε πραγματικά μια τεράστια ευθύνη απέναντι στι γυναίκε του Αφγανιστάν. Δεδομένου ότι υπόθηκε το 2001 και μετά από αυτά που κάναμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το έργο πολυάριθμων ενώσεων στην Ευρώπη και είδαμε την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες και ιδιαίτερα οι γυναικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Έχουμε πραγματικά βαριά ευθύνη σε ό,τι αφορά το μέλλον των γυναικών του Αφγανιστάν. Γιατί δεν έχουν κερδίσει μια ισότητα αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον πολλές από αυτές τις γυναίκες ε, έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που στο παρελθόν ήταν ε, νίκουστες. Συμμετέχω και στην αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Αφγανιστάν και αυτό που λέω είναι ότι μία γυναίκα έχουμε μόνο κυβερνήτρια στο Αφγανιστάν, την κυρία Σοραμπή, που είναι μια εξαιρετική γυναίκα και έχει καταπληκτικό έργο στην επαρχία του Μπαμιάν. Έχουμε τουλάχιστον μία γυναίκα που είναι κυβερνήτη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή και έχει και σημαντικό έργο και στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχει πολλά προσόντα αυτή η γυναίκα. Τουλάχιστον μία γυναίκα να στηρίξουμε αυτή τη γυναίκα ε, στο Αφγανιστάν. Καλύτερα να στηρίξουμε αυτοί παρά τους διεφθαρμένους της Καμπούλ. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Δεν έχω λύσει να, προσ... να προτείνω, αλλά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ κύριε Κιλ Νίλσεν. Το λόγο έχει η κυρία Παπαδοπούλου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Παρακολούθησα με αρκετών ενδιαφέρον τη συζήτηση και ακούστηκαν πολλά και σημαντικά. Ε, προερχόμενοι από την Κύπρο, όπου και εμείς οι Ευρωπαίες γυναίκες της Κύπρου ζούμε σε μια κατάσταση αρκετά παράξενη, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια και το δικό μου νησί είναι μοιρασμένο, ξέρουμε τι είναι οι τραγικές συνέπειες ενός πολέμου. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Είτε γίνεται στο Αφγανιστάν, είτε γίνεται στα Βαλκάνια, είτε γίνεται στην Κύπρο, είτε γίνεται αλλού. Και εκείνο το οποίο ξέρω, γιατί είμαι και εγώ πρόσφυγας, είναι ότι προκαλεί πολύ μεγάλες πληγές που ουδέποτε επουλώνονται. Εγώ μπήκα στην πολιτική ακριβώς γιατί ένιωσα το βάρος της αδικίας ενάντια στη χώρα μου, σαν μια γυναίκα μορφωμένη που μπορεί να ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο και δεν μπορώ να διασχίσω από την πράσινη γραμμή για να επισκεφτώ το πατρικό μου σπίτι που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974. Είδα γυναίκες στη χώρα μου να βιάζονται. Νεαρές γυναίκες, 16-17 χρονών. Να φέρνουν στον κόσμο παιδιά για τα οποία δεν ήταν προϊόν ενός ερώτα. Βιάστηκαν από Τούρκους στρατιώτες. Είδα τη μάνα μου να ξεσπιτώνεται. Και όταν βλέπω γυναίκες στο Αφγανιστάν ή στα Βαλκάνια ή αλλού να υφίστανται την ίδια τραγωδία, πραγματικά συμπάσχω μαζί τους. Γι' αυτό άφησα την επιστήμη μου που ήμουν χημικός για να γίνω πολιτικός και να βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που ανάφερε προηγουμένως μια συνάδελφος, ότι ο πόλεμος δεν είναι λύση και πάντα υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές, είναι το σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταθεί ως θεματοφύλακας αρχών, να μην δέχεται double standards, δεν μπορεί μια χώρα να πηγαίνει να κάνει μια εισβολή και να καταστρέφει και να δικαιώνεται, να μην στυλιτεύεται. Και μιλώ για την Τουρκία. Μιλώ και για το Αφγανιστάν. Εγώ δεν έχω πιστεί για ποιο λόγο να γίνονται επεμβάσεις ή από το ΝΑΤΟ ή από κάποιους. Ο πόλεμος δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν πάντα τρόποι να ενδυναμώσεις τι γυναίκε, να τι στηρίξει, να χρηματοδοτήσει. Και δυστυχώ θα συμφωνήσω με την ομιλήτρια εκεί απέναντι στην άκρη που είπε ότι ο πόλεμο γίνεται για πολιτικού λόγους, για οικονομικού λόγους, για στενά συμφέροντα, εθνικιστικά συμφέροντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι θέμα αν είναι ο άντρα που εξουσιάζει και είναι η γυναίκα συνήθω είναι το θύμα. Και Πιστεύω ότι για να μπορεί να υπάρχει ανατροπή, ναι, θα πρέπει να έχουμε γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταλλάσσει καλές πρακτικές, να στηρίξει με πολλούς πόρους τις γυναίκες όπου και αν βρίσκονται για να μορφωθούν, να έχουν αυτοπεποίθηση, να μπουν στην πολιτική, γιατί η διαφορά της γυναίκας όταν είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ότι θα δουλέψει για μια κουλτούρα ειρήνης δεν θα δουλέψει για τον πόλεμο. Γιατί δεν θέλει να βλέπει τον άντρα τη να σκοτώνεται ή το παιδί τη. Δεν θέλει η ίδια να είναι χείρα. Θέλει να βλέπει γύρω τη την οικογένεια τη να δημιουργεί. Γι' αυτό η δική μου εισήγηση είναι ότι εμεί οι γυναίκε είμαστε αλληλέγγυε. Ανεξάρτητα από ποιο γεωγραφικό μήκο ή πλάτο βρισκόμαστε. Να συνεχίσει ο διάλογο ανάμεσα στι γυναίκε όπου και αν βρίσκονται να στηριχτούν τα γυναικεία κινήματα, ιδίω σε χώρε που βάλλονται από εισβολέ ή από πολέμου. Και οπωσδήποτε να αυξηθούν οι πόροι για να μπορούμε να βλέπουμε τι γυναίκε όταν κατεβαίνουν σε εκστρατείε προεκλογικέ να κερδίζουν, να μην παραμένουν μόνο υποψήφιε. Σε συγκεκριμένε χώρε που υπάρχουν πολεμοί, οι γιατροί του κόσμου πιστεύω κάνουν μια αξιόλογη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι η γυναίκα στο στράτευμα και να είναι στρατιώτης για να στρίξει την άλλη γυναίκα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η γυναίκα να είναι στο στράτευμα. Ο ρόλος της γυναίκας δεν είναι να κρατά όπλο. Ο, ο, ο ρόλος της γυναίκας είναι να χτίζει, να δημιουργεί και όχι να καταστρέφει. Σας ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Δεν βλέπω να υπάρχει καμιά άλλη παρέμβαση. Να δώσω τότε το λόγο στις δύο προσκεκλημένες μας ε, για να ε, κλείσουν τη συζήτηση. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω στα γαλλικά, να απαντήσω. Υποθέτω ότι τα αγγλικά είναι καλύτερα. Δύο παρατηρήσεις. Ε, Υπάρχει μια κυρία που λέγεται Μαρία Μπασία που είναι η πρώτη ε, εισαγγελέα στο ε, δικαστήριο στην Χεράτη. Είναι εκπληκτική γυναίκα. Ε, έχει πετύχει αναγνώριση στι ΗΠΑ. Είναι καταπληκτική γυναίκα πάντω. Την γνώρισα πριν κάποια χρόνια. Δεν μπορώ να απαντήσω στα ελληνικά. Πάντω. η παρουσία των γυναικών στον στους δημόσιους χώρους ε, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, ε, έχουν, έχουν περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών βουλευτών στο Αφγανιστάν από ότι στη Γαλλία, αλλά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν δημοσίω. Ε, δημοσίως. Αυτό που είπε η Κάθριν ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Πρόκειται για γυναίκε που έχουν κοινωνική ισχύ, που μπορούν να μιλούν σε ιδιωτικό χώρο, αλλά θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να μιλάνε και δημοσίως, διότι οι γυναίκες όταν αποκτούν ε, ισχύ τελικά εσωτερικεύουν το πρόβλημα και όπως είδαμε από ε, σημαντικές παρουσίες στο Κανταχάρ οι γυναίκες αυτές εσωτερικεύουν τις, ε, την πολιτική των ανδρών, την πολιτική της κοινότητας που ζουν. Δεν αρκούν τα νούμερα λοιπόν. Μα ενδιαφέρει η πολιτική, μα ενδιαφέρουν οι στατιστικέ, αλλά και η πραγματική γνώση αυτών που γίνονται. Ε, ε, στο Αφγανιστάν έχουμε τρει διαφορετικού νόμου. Έχουμε το Σύνταγμα, όπου τα δικαιώματα των ποινικών αναφέρονται στο άρθρο 27 και τους ε, και, το δικαίωμα να ανοίξει κανεί δική του επιχείρηση στο άρθρο 5. Κατόπιν έχει κανεί τον νόμο Σαρία και κατόπιν έχει και τον παραδοσιακό νόμο που είναι ο πιο ισχυρό. Οι γυναίκε. Ε, ε, θα πρέπει να ληφθούν αυτά λοιπόν υπόψη κατά την εκπαίδευση γυναικών βουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα δώσω τώρα τον λόγο στην Αν Κατρίν Ριεπνίσκη. Παρακαλώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από εμά που να του αρέσει ο πόλεμος. Ούτε και εμένα μου αρέσει, παρότι έχω ε, περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια στο στρατό. Και μερικές φορές, όπως ε, είπε μια ομιλήτρια, πρέπει κανείς να κάνει κάτι. Εγώ η ίδια δεν πήγα στο Αφγανιστάν για να ε, χειροτερέψω τα πράγματα, προσπάθησα να βελτιώσω τα πράγματα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα να θεωρούμε τον πόλεμο ή τους στρατιώτες ως ε, κάτι ε, αποκλειστικά καταστροφικό. Προσπαθούμε να ε, εφαρμόζουμε να επιβάλλουμε την ασφάλεια και πολύ συχνά είναι πολύ σκληρά τα πράγματα και σας διαβεβαιώ ότι πολλά κακά πράγματα θα είχαν γίνει ακόμα χειρότερα αν δεν είχε προσπαθήσει κανείς να παρέμβει. Μπορεί να θεωρείτε ότι είμαι μεροληπτική στο θέμα αυτό, αλλά είναι σημαντικό να ληφθεί αυτό υπόψη. Όλοι μισούμε τον πόλεμο, και εγώ. Υπάρχουν όμως δυνάμεις ασφαλείας ε, που απαιτείται να είναι εκεί. Θα ήθελα επίσης ε, να απαντήσω στην κυρία Κιτ Νίλσον, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Ε, οι Αφγανές γυναίκες ε, είναι τρομοκρατημένες με την ιδέα ότι θα φύγουμε, διότι μας, βλέπουν, μας να αντιμετωπίζουμε τους Ταλιμπάν, να συνομιλούμε μαζί τους και φοβούνται ότι τα πράγματα θα επανέλθουν ε, σε αυτό που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ελπίζω λοιπόν ότι κάποιος θα αγωνιστεί ε, γι' αυτό. Ε, θα χαρώ πολύ αν είστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, να δώσω το λόγο στην κυρία Νικολάη, που είναι η υπεύθυνη συγκήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον αυτό απόγευμα, για, την, για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Θα προσπαθήσω να ψινοψήσω και να ε, σχολιάσω κάπως το θέμα μας. Νομίζω ότι η σεξουαλική βία κατά τις ε, ένοπλες συγκρούσεις, ιδιαίτερα το θέμα του βιασμού, ε, είναι ένα πράγμα που χρησιμοποιείται ως όπλο. Θυμόμαστε τι έγινε στο Κόγκο. Χρειαζόμαστε όμως ε, συγκεκριμένα βήματα. Νομίζω ότι γίνονται πολλά για να καταδικαστεί η κατάσταση και να βελτιωθεί. Σήμερα αναφερθήκαμε στο σχεδικό ψήφισμα. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει πολλά, διότι δυστυχώς δεν έχουν όλες οι χώρες εθνικό σχέδιο δράσης. Σε πολλές χώρες δεν είναι θέμα που να βρίσκεται στην πολιτική ατζέντα. Και ακόμα και αν ε, Έχουμε τελικά ένα σημείο επαφή ε, για τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη πάνω στο θέμα αυτό. Το άλλο θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Από ό,τι κατάλαβα, η, ε, η θέλει να ε, διορίσει ε, ένα άτομο ε, που θα ασχοληθεί με το θέμα της ε, σεξουαλικής βίας. Αυτό αποτελεί πολύ καλή ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε μαζί να οργανώσουμε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι ένα πρόγραμμα εκπαίδευση για αυτού που συμμετέχουν σε ειρηνευτικέ αποστελέ είναι ζωτική σημασία. Δυστυχώ, δεν υπάρχουν ε, πολλές... Ε, δυστυχώς πολλές από τις χώρες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές ε, αποστολές δεν ασχολούνται και με το θέμα του φύλου ώστε να υπάρχει ισορροπία στον τομέα αυτών. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν κάποια προγράμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό όμως δεν ισχύει και σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι ένα πρόβλημα για τα κράτη-μέλη το θέμα αυτό της εκπαίδευσης. Ε, σήμερα δεν ε, αναφερθήκαμε πολύ στο θέμα της καταδίκης. Ακόμα και αν υπάρχει τεράστιος αριθμός υποθέσεων, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, σχετικών καταδικών. για τη Βοσνία είχαν αναφερθεί 50.000 υποθέσεις βιασμού. σε, επίπεδο εθνικής δικαιοσύνη όμως ε, υπήρχαν μόνο 12 ε, υποθέσεις ποινική δίωξης. Ίσως είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη δίωξη στις περιπτώσεις ε, βιασμού. Και ίσως να πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, και σε θέματα φυλετικής ε, ισορροπίας. Διότι στα πανεπιστήμια, στις νομικές σχολές, όταν, προετοιμάζεται, όταν προετοιμάζονται οι φοιτητέ για τέτοια θέματα, το θέμα του φύλου δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δυστυχώς δεν είναι πολλοί οι εισαγγελείς ή οι δικαστές που να μπορούν να ανταποκριθούν ε, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον φίλο. Και ο ε, στιγματισμός ε, είναι μια συνέπεια της σεξουαλικής ε, βίας. Και τέλος, πιστεύω ότι μαζί θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τεθεί το θέμα πια στην ημερήσια διάταξη και θα είναι επιτυχής η δράση μας μόνο εάν ε, αποκτήσουν περισσότερη δύναμη, περισσότερη ισχύ οι γυναίκες. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα κλειδί στην όλη υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νικολάη. Είπα στην αρχή της ακρόασής μας ότι προσβλέπουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα και ε, διαπιστώνω τώρα ότι ήταν εξαιρετικά ε, ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση. Ακούσαμε διάφορες ε, εμπειρίες των προσκεκλημένων μας Ακούσαμε πυρογνώμονα για τον αφοπλισμό, ακούσαμε ε, ανθρώπους που ασχολούνται με θέματα ισότητας ε, στην άμυνα και ακούσαμε τις εμπειρίες ε, γυναικών στην πράξη. αυτές ε, οι διάφορες ε, δεξιότητες ε, των γυναικών που ήταν σήμερα προσκεκλημένες μας βοήθησαν να αποκτήσουμε μία πολύπλευρη εικόνα σήμερα το θέμα μας ήταν η συμμετοχή των γυναικών κατά τις συζητήσεις αφοπλισμού, κατά την επανικοδόμηση και την ε, συμμετοχή τους ε, στην πραγματικότητα στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο να υπάρχουν γυναίκε στι οποίε να μπορεί να απευθυνθεί κανεί να ζητήσει βοήθεια. Μάθαμε λοιπόν πολλά πράγματα. Ε, ελπίζω λοιπόν τώρα ότι τις γνώσεις αυτές που αποκτήσαμε θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να σημειώσουμε μαζί πρόοδο. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τις προσκεκλημένες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ε, ευχαριστώ την ε, Γραμματεία. Η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά και τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή μας στις 9 ακριβώς σε τούτη την αίθουσα. Σας περιμένω λοιπόν αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.